Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να καθίσετε. Αρχίζει η συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Είναι πάρα πολύ σημαντική. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Θα περάσουμε αμέσως στην ημερήσια διάταξη. Δεν υπάρχουν παρατηρήσεις για τη σημερινή ημερήσια διάταξη, δεν βλέπω τίποτα. Οι διερμηνεί σα πληροφορούν με τα λύπη ότι συνεχίζεται η εργασιακή διαμάχη με τη διοίκηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τι νέε συνθήκε εργασία που αποτέλεσε το αντικείμενο προειδοποίηση για απεργιακή κινητοποίηση. Η ποιότητα τη διερμηνία κινδυνεύει για του Ευρωβουλευτέ και του Ευρωπαίου πολίτε. Δυστυχώ, λόγω τη εργασιακή διαμάχη, η διερμηνία θα σταματήσει στι 10.30 ακριβώ, όπω προβλέπει το πρόγραμμα τη συνεδρίαση. Λοιπόν, ο κύριος Επίτροπος θα μας παρουσιάσει τρεις ε, προτάσεις. Είναι η πρόταση 392, νομοθετική πρόταση που, που την έχει ήδη εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επίτροπη. Καλωσορίζουμε τον Επίτροπο στο Κοινοβούλιο. Το Κοινοβούλιο έχει ολοκληρώσει τις εργασίες του και εδώ αναφέρομαι στην έκθεση Dorfman η οποία εγκρίθηκε στις 20 Μαΐου. Λοιπόν, ακολουθούμε τη διαδικασία, την ημερήσια διάταξη και όταν έχουμε ε, κάποια προβλήματα που έχουν σχέση με την νομοθεσία θα τα δούμε μετά την παρουσίαση του εγγράφου. Ε, θα πρέπει να δούμε λοιπόν ε, τι συνέχεια θα δώσουμε. Στα διάφορα θέματα θα ορίσουμε εισηγητές και θα κάνουμε συζητήσεις, διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες και ειδικούς και πιστεύω ότι Ξέρουμε όλοι ότι βρισκόμαστε στο τέλος της θητείας, οπότε ε, είναι πάρα πολύ γνωστές οι προθεσμίες και πάρα πολύ σφιχτά τα χρονοδιαγράμματα. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε στο υπόλοιπο που μας απομένει της θητείας να φέρουμε σε πέρας, αίσιο πέρας όλα αυτά που μας απομένουν. Ε, τα νομοθετικά εννοώ. Πριν σας δώσω το λόγο κύριε Επίτροπε, θα ήθελα και πάλι να σας ε, παρουσιάσω το χρονοδιάγραμμα μάλλον όχι την, την, την ε, πορεία των εργασιών. Οι συντονιστέ θα μιλήσουν δύο λεπτά, μετά θα απαντήσετε εσεί κύριε Επίτροπε, μετά οι υπόλοιποι ε, συνάδελφοι ένα λεπτό θα ξανά και προτεραιότητα θα έχουν ε, οι βουλευτές που λαμβάνουν το λόγο για την αλληλεία. Παρακαλώ, έχετε το... Thank you very uh, Uh, ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη στην Επιτροπή για την μικρή μου καθυστέρηση. Κανείς ποτέ δεν μπορεί να κάνει προβλέψεις ε, στην Γαλλία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που οργανώσατε αυτή τη συνάντηση στην οποία θα γίνει μια ανταλλαγή απόψεων με την πρόταση της Επιτροπής για την ΚΑΠ. Θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας τον εισηγητή για το, που έκανε την έκθεση για το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω μια πάρα πολύ επικοδομητική και χρήσιμη έκθεση, μια έκθεση την οποία ψηφίσατε και στην Επιτροπή και στην Ολομέλη και συμβάλλει τα μάλλα στη εργασία μας. Θα επανέλθω στο θέμα αυτό αργότερα. Βεβαίω, η πρόταση της Επιτροπής αποτελεί το τέλος της φάσης 1 της διαδικασία και την απαρχή μια καινούρια φάσης της διαθεσμική. Θα συμφωνείτε ότι η πρόταση της Επιτροπής αποτελεί τουλάχιστον μια καλή βάση κίνησης και εργαζόμενοι επικοδομητικά θα μπορούσαμε να την βελτιώσουμε προς το όφελο ε, των αγροτών. Και εγώ μπορώ να σας διαβεβαίωσω ότι είμαι στη διάθεσή σα για να λάβω υπόψη με οποιαδήποτε υπόδειξη θα έτεινε στη βελτίωση της πρόταση. Πρόκειται για μια ρεαλιστική, εξισορροπημένη και φιλόδοξη προσπάθεια και έχει σχέση με τόσο δεσμευτήκαμε να κάνουμε τον Νοέμβριο. Έχει σχέση με το πλαίσιο για μια περισσότερο βιώσιμη κοινή αγροτική πολιτική βρισκόμαστε αντιμέτωποι με νέες προκλήσεις σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο. Θεωρώ ότι είναι καθήκον μου να δώσω στους αγρότες την βεβαιότητα και την δυνατότητα να προβλέψουν λαμβάνοντας υπόψη σε επενδύσεις που θα πρέπει να κάνουν. Η πρόταση αυτή γίνεται με βάση αυτό το πνεύμα και νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί κίνδυνοι του να μην επιτευχθεί μια συμφωνία. Μίλησα για τις προκλήσεις σε σχέση με το προπολογισμό και φαίνεται ότι είναι σκόπιμο να περάσουμε σε θέματα ουσίας να πω κάτι για μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις. Σε εννέα μήνες από τώρα το Ενωμένο Βασίλειο, ένας από τους ε, που συμβάλλουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πείσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό θα πείσει ένα κενό στον προπολογισμό. Αυτό είναι γνωστό σε όλους. Αυτό γίνεται παράλληλα με την σύμφωνη γνώμη των μελών ότι θα πρέπει να τεθούν άλλες προτεραιότητες σε ό,τι αφορά την μετανάστευση και την ε, προάσπιση των Ευρωπαίων. Λαμβάνοντας λοιπόν όλα αυτά τα θέματα μαζί και τη απουσία ομοφωνίας σε ό,τι αφορά την αύξηση των εισφορών στον προπολογισμό, η Επιτροπή έχει θέσει μια νέα πρόταξη, πρόταση γιατί θα μπορούσε να προκύψει ένα έλλειμμα. Σε αυτό το πλαίσιο, η πρόταση της Επιτροπής για μείωση στον προλογισμό κατά λιγότερο από 5% και 2-12% σταθερές τιμές είναι κάτι που θα πρέπει να εξεταστεί για λόγους ε, διαφάνειας ε, η Επιτροπή υπέβαλε την πρότασή της και στις δύο τιμές και βρίσκονται ενώπιόν σας για να τις δείτε. Είδα και μερικές άλλες ε, αναλύσεις που δείχνουν ότι υπάρχει κάποια έλλειψη τιμιότητα στον τρόπο τον οποίο παρουσιάζονται τα δεδομένα. Δεν πιστεύω όμως ότι δεν καταλαβαίνω αυτή την εναλλακτική ανάλυση και δεν καταλαβαίνω ποια βάση ξεκινάει. Συνεπώς δεν βρίσκομαι για να ξεκινήσω μια ακαδημαϊκή συζήτηση σχετικά με το πώς μετράμε και συγκρίνουμε τους πολιτείς προϋπολογισμούς. Οι γεωργοί ξέρουν πάρα πολύ καλά πώς συγκρίνουν τα στοιχεία μεταξύ του 20 και του 21. Αυτό που μετράει είναι το τελικό αποτέλεσμα για τον γεωργό. Σε μια προσπάθεια διαφάνειας, σε μια προσπάθεια να βοηθήσουμε Συντάξαμε ένα λεπτομερές έγγραφο εργασίας που παρέχει τεχνικές εξηγήσεις συμπεριλαμβάνοντας θέμα που αφορούν την αιτήσια ανάλυση και παρεμφερή θέματα. Οι υπηρεσίες μου θα συνεχίσουν να είναι στη διάθεσή σας αν χρειάζεστε οποιαδήποτε διευκρίνηση, οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Ο προπολογισμό αποτελεί αποτέλεσμα των περιστάσεων Άκουσα με προσοχή τις αντιδράσεις ορισμένων κρατών μελών, ιδιαίτερα όσες ακούστηκαν στην ε, Σόφια, αλλά άκουσα και τις παρατηρήσεις των Ευρωβουλευτών ό,τι αφορά την καταλληλότητα του προπολογισμού. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι αν φτάσουν περισσότερα χρήματα, εγώ δεν θα σταθώ εμπόδιο. Ούτε εσείς, ούτε κανένας άλλος αλλά θα πρέπει να υπάρξει σύμφωνη γνώμη όλων προκειμένου να συμβεί κάτι τέτοιο. Ε, υπήρξαν ορισμένοι που είπαν ότι θα πρέπει να διατηρηθεί ο υπάρχον προπολογισμό. Εναπόκειται τώρα στα κράτη-μέλη και σε άλλους να αποφασίσουν πώς θα επιτευχθεί αυτό. Τα τελευταία αποτελέσματα θα ε, ε, εξαρτούν από τα κράτη. Εγώ θα κάνω κάθε προσπάθεια για να βελτιώσω τα πράγματα στον κλάδο της γεωργίας. Στην πολιτική πρέπει να κάνουμε επιλογές, κυρίως όταν λείπουν τα χρήματα. Και αυτό το τόνισα από την αρχή της ε, θητείας μου. Έχω την ε, ευτυχία να συναντώμε συχνά με πολλούς από εσά και νομίζω ότι θα μπορούμε να πούμε ότι οι αδυναμίες που έχουμε εντοπίσει από κοινού συνέβαλαν στις επιλογές που κάναμε και η βασική επιλογή είναι να δώσουμε προτεραιότητα τη στήριξη του εισοδήματο των γεωργών. Θεωρώντα ότι αυτό απαιτείται προκειμένου να μπορέσουν οι γεωργοί να τρέφουν ελπίδες βιωσιμότητας, οι ίδιοι και οι οικογένειε τους. Γιατί όταν συγκρίνεται τη γεωργία από, με άλλους κλάδους το 46% των εσόδων προέρχεται από άμεσες ε, πληρωμές. Το υπόλοιπο προέρχεται από την αγορά. Έχουμε διατηρήσει την εξωτερική σύγκληση και αυτό σημαίνει οι περισσότερες φορές. Βεβαίως, ε, ορισμένοι θα ήθελαν ένα πιο φιλόδοξο πρόγραμμα. Αυτό χρειάζεται περισσότερα χρήματα. Έχω την βεβαιότητα ότι κανένα ε, δεν λέει ότι θα πρέπει να γίνουν περικοπές στο προπολογισμό. Ε, ελπίζω να έχουμε περισσότερα χρήματα για να επιτευχθεί περισσότερη πρόοδος. Προκειμένου να υπάρχει μια δικαιότερη κατανομή των πληρωμών και για να βοηθήσουμε το, ε, τους γεωργούς που είναι σπονδυλική στήλη Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής η Επιτροπή υπέβαλε προτάσεις. Καταρχάς, ένα υποχρεωτικό κάπινγκ, έτσι ώστε δεν θα επηρεάσει τα πράγματα την απασχόληση. Οι χώρες μένει μπορούν να θέσουν να κάνουν μεταξύ 60 και 1.000 ευρώ. Ελπίζουμε ε, και τα έσοδα θα διανεμηθούν σε κάθε χώρα μέλος. Δεύτερον, τα κράτη-μέλη θα μπορέσουν να δώσουν ένα επάπαξ ποσό στα μακρά αγροκτήματα. Πολύ πιο εύκολο από το να κάνουμε κάτι άλλο. Τρίτον, σε ό,τι αφορά την εσωτερική σύγκληση στο τέλος της περίοδου του MFS καμία πληρωμή ένα εκτάριο μπορεί να είναι λιγότερο από 70% του βασικού ε, που δίνεται για κάθε κράτο μέλος. Στα πλαίσια της ε, συγχρηματοδότησης μέσω όλων των ταμείων θεωρήσαμε ότι ήταν ε, αναγκαίο να θέσουμε και πάλι το θέμα της συγχρηματοδότησης. η Ευρωπαϊκή Ένωση αναλαμβάνει ένα μέρος της χρηματοδότησης στο δεύτερο πυλώνα σε 15,7%. Ε, ε, ε, αυτό το κάναμε λόγω της δυνατότητας από τα κράτη-μέλη στον πυλώνα 2 να καλύψουν αυτό το κενό μεταφέροντας από το 2 στο 1. Έχουν επιλογές. Οι χώρε μέλη έχουν αυτέ τι ε, δυνατότητες αν θεωρούν ότι ο πυλώνα 2 είναι η προτεραιότητά τους και δεν είναι το ένα. Είχαμε την ε, ευκαιρία να διατηρήσουμε την ε, πολιτική προσανατολισμένη προς την αγορά. Αυτό είναι σημαντικό. Όχι για λόγους ιδεολογίας ή για διεθνή, λόγω διεθνών κανόνων. Γιατί χωρίς κάτι τέτοιο η οικονομική χωρις κατι τετοιο οικονομικη βιωσιμοτητα θα αρχίσει να διακυβεύεται. Θα πρέπει να δούμε πώς θα στηρίξουμε τον προσανατολισμό στην αγορά Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της ενδυνάμωσης της θέσης των γεωργών, βασίζουμε στι αλλαγές που κάνατε ήδη στον κανονισμό και στην πρόταση της Επιτροπής η μελλοντική ΚΑΠ θα παράγει δυνατότητες υποστήριξης των οργανώσεων των παραγωγών για κοινέ δράσεις μείωση του κόστους εμπορίας και μείωση της πατάλης τροφίμων. Αυτό θα γίνει με βάση δύο προγράμματα και θα ε, είναι ανοιχτό για όλους τους τομείς της γεωργίας. Όπως μπορείτε να δείτε, θέλουμε να πέσουμε, ε, να δημιουργήσουμε νέες ευκαιρίες και θέλουμε να ενδυναμώσουμε το ρόλο των γεωργών στην τροφική Θα δοθεί πάρα από το 3% του πυλώνα 1 και ελπίζουμε να μπορέσουμε να το κάνουμε. Κύριε Πρόεδρε, δεν πρέπει να σας επλήξει το γεγονός ότι ε, υπάρχει πρόταση για το περιβάλλον και το κλίμα αυτό. Το είδαμε στην ανακοίνωση του Νοεμβρίου. Ήδη αναφέρεται στην Συμφωνία του Παρισίου, δηλαδή οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης για το 2025. Ξέρω ότι κοιτάζετε τις ε, διάφορες ε, μελέτες και ξέρω ότι γνωρίζετε ότι οι πολίτες αποδίδουν μεγάλη σημασία στα γεωργικά προϊόντα. Θα πρέπει να στηρίξουμε όμως ε, τους γεωργούς. Και ένας από τους βασικούς στόχους του μέλλοντος του ΚΑΠ είναι να υπάρξει περιβαλλοντική δράση. Υπάρχουν τρεις στόχοι εδώ σε ό,τι αφορά την νομοθεσία και αυτό δείχνει την περιβαλλοντική σημασία της πολιτικής. Ακούσαμε και απαντήσαμε στους ε, ε, επικριτές της πράσινης αρχιτεκτονικής της ΚΑΠ. Αποφασίσαμε να διακόψουμε τη, και να την αντικαταστήσουμε με μέτρα που είναι περισσότερο κατάλληλα. Ενδυνάμωση δηλαδή του περιβάλλοντος για τις άμεσες πληρωμές το 30% της χρηματοδότησης θα πρέπει να αφορά μέτρα βιοπικιλότητας, αποκλείοντας πληρωμές ESCP στον πυλώνα 2, ελαστικότητα μετακίνησης μεταξύ των πυλώνων και αν οι χώρες μέλη θέλουν να έχουν τη δυνατότητα μπορούν να το κάνουν με ένα επιπλέον 15% χωρίς να υπάρχει ανάγκη για ε, εθνική χρηματοδότηση. Επίσης δώσαμε ευκαιρίες για τις χώρες μέλη ε, για σχήματα στο πρόγραμμα. Ένα που θα πάνε ε, πέρα από τις ε, προϋποθέσεις. Θα υπάρξουν δηλαδή επιμέτρο αποφάσεις. Οι δράσεις αυτές της ΚΑΠ θα συμβάλλουν στο 40% του προπολογισμού σε ό,τι αφορά το κλίμα. Κύριε Πρόεδρε, για τρία χρόνια προσπαθήσαμε να απλοποιήσουμε την ΚΑΠΑ. Πάνω από 100 μέτρα ψηφίστηκαν τα τελευταία χρόνια. Βεβαίω θα πρέπει να κάνουμε περισσότερο. Η πολιτική αυτή αποτέλεσε αντικείμενο κριτικής λόγω το, της πολυπλοκότητάς της. Δύο πτυχές του νέου μοντέλου θα εξασφαλίσουν απλοποίηση. Το πρώτο είναι ότι οι κανόνες ε, θα συνδέονται περισσότερο με την πραγματικότητα των δικαιούχων, οι χώρες μέλη θα επιλέγουν τα μέτρα και θα αποφασίζουν τους κανόνες, όπως τα κριτήρια επιλεξιμότητας που θα βασίζονται σε ένα πρόγραμμα της ΚΑΠ. Θα υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια, μεγαλύτερη λογοδοσία, μεγαλύτερη κατανόηση. Οι κανόνες μπορεί να ε, οριστούν με καλύτερο τρόπο. Η δεύτερη πτυχή του μοντέλου αυτού που θα οδηγεί σε απλοποίηση είναι ότι αυτό που θα μας απασχολήσει πρωτίστως είναι τα αποτελέσματα και οι επιδόσεις. Θα μειωθούν οι έλεγχοι και θα περιοριστούν σε γενικές ε, γραμμές και όχι στα προπετούμενα για τους ε, γεωργούς. Νομίζω ότι αυτό θα βρει σύμφωνο τους γεωργούς. Η χρήση νέων τεχνολογιών θα αυτοματοποιήσει και θα επιταχύνει πολλές από τις διαδικασίες. Οι γεωργοί θα έχουν βελτιωμένη πρόσβαση στη συμβουλευτική και θα υπάρξει μείωση της γραφειοκρατίας. Υπάρχει ε, και η τεχνολογία ε, του Κοπέρνικου η οποία δίχως ε, θάλο θα βοηθήσει τον έλεγχο και τη λειτουργία της ΚΑΠΑ. Θα ανακύψουν πάρα πολλά πλεονεκτήματα από τους γεωργούς στο μέλλον θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν ε, ένα σύστημα μακρινής παρακολουθήσης των γεωρικών δραστηριοτήτων. Αυτό θα διασφαλίσει με σχετικά χαμηλό κόστος τη διαθωσιμότητα ε, συγκρίσιμων ευρωπαϊκών δεδομένων ε, για στόχους διαχείρισης της πολιτικής, ότι πρόκειται για την επιστήκη ασφάλεια, για το κλίμα, για το περιβάλλον κτλ. Αυτό θα γίνει στο μέτρο του δυνατού και θα αντικαταστήσει τις κλασικές μεθόδους ελέγχου, όπως τους ελέγχους επιτόπου που θα μειώσουν το διοικητικό άχθος και θα μειώσουν πιθανότητα το άχθος του ελέγχου επί των Γιώργο. Μια τέτοια προσέγγιση θα βοηθήσει τους γεωργούς να μειώσουν το χρόνο και την πολυπλοκότητα για να υποβάλουν τις αιτήσει τους και κάποια κράτη-μέλη μάλιστα σκέφτονται να αναπτύξουν ε, ένα πρόσκοπτο σύστημα υποβολής καταγγελιών. Ε, θα μπορέσουν έτσι λοιπόν οι αγρότες ε, να συμμετέχουν και να μπορούν να ελέγχουν τις απαιτήσει επιλεξιμότητας. Αυτό σημαίνει ότι θα χρησιμοποιείται λιγότερος χρόνος και θα μπορούν να χρησιμοποιούνται πιο εύκολα οι όροι επιλεξιμότητας. Θα επωφεληθούν οι γεωργοί από τις νέες τεχνολογίες θα μπορούν να διαχειριστούν καλύτερα τις εκμεταλλεύσεις τους ε, και θα έχουμε και αυτό με τη καταγραφή των δραστηριοτήτων, κάτι που θα μειώσει την ε, ε, γραφειοκρατία. Θα υπάρχει και πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλο για τα κράτη-μέλη, αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων ε, ε, θα μπορεί να ε, εφαρμόσει καλύτερα τα κριτήρια επιλεξιμότητας, θα έχουμε μείωση του κόστου με τις φυσικές επιθεωρήσεις επιτόπου και θα έχουμε πιο επικαιροποιημένα στοιχεία λόγω της διαδικασίας επισκόπηση, η ανάλυση των γεωλογικών ειδικών δεδομένων και των μετρήσεων σίγουρα ζητείται πάρα πολύ από ανθρώπους που εργάζονται στον τομέα. Και επίσης η ε, εφαρμογή ε, για τον γεωγραφικό χώρο είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για να αποφευχθούν τα λάθη ε, στις δηλώσεις και να αποφευχθούν επιβολές κυρώσεων στους γεωργούς και θα γίνει μετά το 2020 ο κύριος τρόπος υποβολής των δηλώσεων. Τα κράτη-μέλη θα μπορούν εκ των προτέρων να συμπληρώνουν την αίτηση ε, με επικαιροποιημένες και αξιόπιστες πληροφορίες. Έτσι λοιπόν θα υπάρχει ένα σύστημα που σχεδόν δεν θα κατατίθονται παράπονα και θα ζητείται απλώ να επιβεβαιώσει ο Γιώργος τη δήλωση που θα υποβάλει η δίκηση. Αυτή είναι μεγάλη αλλαγή προς το να βοηθήσουμε τους Γιωργούς και η δίκηση βοηθά τον Γιώργο. Ένα ερώτημα που θέλω να θέσω έχει να κάνει με την καρδιά της ΚΑΠ. Είναι ένα ε, θέμα της ε, κινησφής. Όλα τα διάφορα στοιχεία που ανέφερα θα συνεισφέρουν έτσι ώστε να παραμείνει η ΚΑΠ μια πραγματική κοινή πολιτική με ένα κεφαλαίο ΚΑΠΑ. Θα βασίζεται στη σωστή ισορροπία μεταξύ αυτής της κοινή φύσης και της απαραίτητης ευελιξίας για τα κράτη-μέλη και μάλιστα και σήμερα έχουν ευελιξία για να απαντήσουν αποτελεσματικά στις ε, τοπικές συνθήκες. Ε, πολλές φορές έχουμε πει ότι πρέπει να απομακρυνθούμε από την προσέγγιση ότι ένα μέγεθος κάνει σε όλους. Ε, θα πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο στις επιδόσεις. Μπορούμε να μειώσουμε το διοικητικό όφελος για τους γεωργούς χωρίς να υποχωρούμε από την κλίση που έχει η κοινή αγροτική πολιτική. Αυτή είναι η ισορροπία που επιζητούμε και σας καλώ να συνεργαστούμε για να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε καλά αποτελέσματα για τους γεωργούς αλλά ε, και για τους ε, πολίτες ε, που θέλουν να πετύχουμε τους στόχους μας όπως είναι η προστασία του περιβάλλοντος, η κοινωνική συνοχή και η πιστιστική ασφάλεια. Θέλω να σας πω ποιες δικλείδες ασφαλείας προτείνουμε ε, για να μην έχουμε ε, επανεθνικοποίηση. Η νομοθεσία θα συμπεριλάβει τους κοινού στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις βασικές απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, που θα εφαρμόζεται στα είδη των παρεμβάσεων, καθώς και πολλά κοινά στοιχεία. Το σχέδιο της έγκρισης για τα στρατηγικά σχέδια ΚΑΠ θα περιλαμβάνει μια ολική αξιολόγηση της σύστασης και της συνεκτικότητας της πολιτικής σε σχέση με τους κύριους στόχους. Και τα κράτη-μέλη λοιπόν θα υποστηρίζονται οικονομικά αλλά και με άλλου τρόπου από την Κομισιόν στην προετοιμασία των σχεδίων αυτών. Η εποβολή εκτίσεων εκθέσεων για τις επιδόσεις ε, θα μας ε, επιτρέψει να δούμε ποιες είναι οι επιδόσεις ε, των κρατών μελών και η Κομισιόν θα μπορέσει να έχει μια διορθωτική δράση κατάλληλη όπως κάνουμε σήμερα Επίσης, θα ζητάμε τα κράτη-μέλη να καταρτήσουν σχέδια πληρωμών θα υπάρχουν κατάλληλε απαιτήσει αξιολόγηση, θα πρέπει να σχεδιαστούν για να επιτρέψουμε έγκαιρη αξιολόγηση των επιδόσεων τη πολιτική. Και ενώ ένα κράτο μέλο θα είναι υπεύθυνο για την αξιολόγηση των στρατηγικών σχεδίων, η Κομισιόν θα, θα παρουσιάσει μια τελική έκθεση για τα τελικά αποτελέσματα της... Ε, των επιδόσεων μετά από τα τρία έτη τη εφαρμογή του σχεδίου. Έτσι, λοιπόν, ε, θα ε, έχουμε ένα μέτρο κατά της ε, πανεθνικοποίησης. Εγώ κάνω το ίδιο εδώ. Χαίρομαι που ε, θα έχουμε αποφύγει κάτι τέτοιο. Στις αρχές ανέφερα την έκθεση Dorfman και την σημαντική συνεισφορά της έκθεσης αυτής. Μετά την υιοθέτηση στην Ολομέλεια, οι υπηρεσίες μου ανάλυσαν προσεκτικά την πρόταση προκειμένου να δουν σε ποιο επίπεδο μπορούμε να συμφωνήσουμε και ποιες είναι οι διαφωνίες ε, που υπάρχουν σε σχέση με την πρόταση της Κομισιόν. Το συμπέρασμά μου είναι ότι το 90% των συστάσεων της ε, έκθεσης ε, και οι παρατηρήσεις ή τα λοιπά σχόλια λαμβάνονται υπόψη στην πρόταση της Κομισιόν, στις προτάσεις της Κομισιόν. Επομένως, το βασικό, ο βασικός τομέας διαφορών αν θέλει Ερικ μπορούμε να το δούμε, αλλά περί αυτού πρόκειται. Το κύριο θεματική των διαφορών έχει να κάνει με τα χρήματα, με τον προπολογισμό. Και ήδη αναφέρθηκα σε αυτό. Σε σχέση με τις ε, νέε σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, τα κράτη-μέλη της Περιφερείας και τους γεωργού, έχουμε επαναλάβει τις δεσμεύσεις μα ε, στι συνθήκε. έχουμε τονίσει τη σημασία, το ρόλο που παίζουν οι μικρομεσαίοι γεωργοί, έχουμε διασφαλίσει ότι τα κράτη-μέλη θα έχουν επαρκή ευελιξία μέσα σε ένα κοινό πλαίσιο ευρωπαϊκών κανόνων. Είναι πολύ γνώριμη αυτή η φράση, Μόλι την ψηφίσατε. Επίση έχουμε αναγνωρίσει το πρόβλημα του κανονιστικού υπερθυματισμού στα κράτη-μέλη. Επίση, ε, προβλέπουμε πώ θα επιλύσουμε το θέμα των καθυστερημένων πληρωμών. Έχουμε διατηρήσει το καθεστώ για του μικρού γεωργού. Έχουμε αντιμετωπίσει τη δυσκολία στον ορισμό του ενεργού γεωργού και έχουμε διατηρήσει την έννοια ε, του γεωργού ω μερική απασχόληση για να έχουμε μια βιώσιμη και δίκαιη ΚΑΠ ε, η οποία θα φροντίζει το περιβάλλον και του γεωργού. Έχουμε κρατήσει τη δομή των δύο πυλώνων. Θα έχουμε πληρωμές που χρηματοδοτούνται πλήρως από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υποστηρίζουμε την έρευνα και την ανάπτυξη μέσω του ορίζοντα 2020 με πρόσθετα 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχουμε ε, σε ευαίσθητες περιοχές και σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς προστατεύσει τους γεωργούς. Επίσης, θέτουμε στο στόχο τις οικογενειακές επιχειρήσεις. Ε, διατηρήσαμε το ΣΑΠ στην ενιαία ενίσχυση και διατηρούμε την ερεσιμότητα σε τομείς ε, όπως ε, δημόσια αγαθά και περιβαλλοντικά παραδοτέα. Επίσης έχουμε διαφυλάξει ε, το θέμα της βελτίωσης ε, της εσωτερικής σύγκλησης και έχουμε διτηρήσει και την πρωτοβουλία Smart Village. Επίσης έχουμε διατηρήσει το πλαίσιο της κοινή οργάνωσης αγοράς στον πυλώνα 1. Επιτρέψαμε την απλούστευση των νομικών απαιτήσεων και μεγαλύτερη ευελιξία για τα κράτη-μέλη για να σχεδιάσουν τα δικά τους εργαλεία διαχείρισης κινδύνου και έχουμε ένα κεφάλαιο με έκτακτα μέτρα στον κανονισμό της ΚΟΑ. Και τέλος, σε σχέση με μια διαφανή διαδικασία ε, λήψης αποφάσεων, συμφωνήσαμε με το να έχουμε ένα κοινό ισχυρό πλαίσιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσα στη διαδικασία της συναπόφασης. Φυσικά πρέπει να γίνει μεγάλη πρόοδος μέχρι τα τέλη της σημερινής ε, θητείας, της τρέχουσας θητείας. Αναγνωρίζουμε τον κριτικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν ε, οι τεχνολογίες του χώρου και προβλέπουμε καλύτερη ολοκλήρωση της κυκλικής οικονομίας σε ό,τι αφορά την αρχιτεκτονική του πρασινίσματος έχουμε προτείνει με ενισχυμένη και απλουστευμένη αιρεσιμότητα για τον πυλώνα 1 που θα είναι υποχρεωτική και έχουμε ένα νέο απλουστευμένο καθεστώς με κανόνες που θα πάει πέρα από αυτό, το εξήγησα ήδη ε, και έχουμε ε, γεωπεριβαλλοντικά εκούσια μέτρα στον πυλώνα 2. Επίσης, βλέπουμε έναν πολύ μεγάλο ρόλο για την καινοτομία και την κατάρτιση στις μικρές και μεσές εκμεταλλεύσεις. Έχουμε αναφέρει ε, στην έκθεσή σας, ε, συγγνώμη, κάνουμε μια αναφορά και στο ε, σχέδιο που αναφέρεται στην έκθεσή σας σε σχέση με τις ενισχύσεις. Έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα τα οποία ήδη ψηφίσατε και έχουμε κοινέ απόψεις μεταξύ ημών και της Κομισιόν και εγώ πιστεύω ότι υπάρχει μια βάση για να συνεργαστούμε. Θέλω να ολοκληρώσω τώρα, Πρόεδρε, να πω ότι ε, τι ε, λεπτομέρειε τη πρόταση θα τις συζητήσουμε τι επόμενε εβδομάδε ε, και μήνε ε, και εγώ και οι υπηρεσίε μου. Φυσικά είμαστε διαθέσιμοι να συζητήσουμε λεπτομερώς. Φυσικά και πολιτικά μπορούμε να συζητήσουμε για όλες τις πτυχές τη πρόταση. Θέλουμε να αντιμετωπίσουμε, να επιλύσουμε κάποια από τα κύρια πολιτικά ζητήματα που σχετίζονται με τι προτάσει που εσεί και εγώ έχουμε υποβάλει και να απαντήσουμε σε κάποιε πρώιμε αντιδράσει. Οι προτάσει Κομισιόν είναι το σημείο αφετηρία και αποτελούν ένα καλό σύστημα απλούστευση και ξεχρονισμού τη πολιτική βάσει των δικών σα εκθέσεων και όσων είδαμε και στα κράτη-μέλη. Από τους Υπουργού Γεωργίας ε, θα ήθελα να σας καλωσορίσω σε επικοδομητική συνεισφορά. Η εμπειρογνωμοσύνη που έχετε είναι πολύ σημαντική για να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα για τους Γεωργούς και ελπίζω να μπορέσουμε να το κάνουμε με ένα συνεργατικό τρόπο τους επόμενους μήνες και να βελτιώσουμε την πρόταση όπου πιστεύουμε ότι μπορούμε να το πράξουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρο. Λοιπόν, κύριε και κύριοι, έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, διότι ο κύριο Επίτροπο μίλησε περισσότερο από ό,τι συνηθίζεται και 40 συνάδελφοι ζητούν το λόγο. Δύο λεπτά ο κάθε συντονιστής και μετά οι υπόλοιποι, αφού ακούσουμε τι απαντήσει του κύριου Επιτρόπου και οι βουλευτέ, εκτό από του συντονιστέ, θα έχετε ένα λεπτό. Έκαστος και κάστη. Παρακαλώ να τηρείτε του χρόνου σας. Λοιπόν, μην αρχίσετε με τι ευχαριστίες. Θα σα φάει το χρόνο. Όλοι μαζί τον ευχαριστούμε τον Επίτροπο. Λοιπόν, 15 δεύτερα πριν λήξει ο χρόνο σα θα σηκώνω σφυρί. Ο κύριο Ντές. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε. Ωραία αυτά που λέτε, αλλά δεν με πείθετε. Στη δεκαετία του 90, ένας ε, ε, ε, πρόσωπος ε, των Γεωργών ορίστηκε επιχειρηματίας της χρονιάς γιατί είχε κάνει κάτι τρομερές εφευρέσεις σε αμελτικές μηχανές και τα λοιπά και γεωργικές εκμεταλλεύσεις. τάζεται λαγού με πέτρα χίλια. Μιλάτε για μείωση της γραφειοκρατίας. Εγώ φοβάμαι ότι τελικά θα έχουμε περισσότερη γραφειοκρατία και όχι λιγότερη. Ειδικά ως Γερμανός βουλευτός ξέρω ότι αν είναι αρμόδια η δική μου χώρα, από τις 27 χώρες θα έχουμε την πιο γραφειοκρατική ε, ρύθμιση. Γιατί καμιά φορά οι ευρωπαϊκές ρυθμίσεις είναι καλύτερες από τις εθνικές και δεν μου αρέσει αυτό. Το Σαββατοκύριακο μίλησα με νέους αγρότες και τους παρουσίασα τις προτάσεις σας γενικά και πολλοί μου είπαν ότι αν ισχύσουν αυτά στο μέλλον σιγά μην παραμείνω εγώ αγρότης. Ε, και ε, πολύ αγωνίο εκεί που βάζουμε πολλά λεφτά στο δεύτερο πυλώνα, όπως στην πατρίδα μου τη Βαβαρία, δεν θα μπορέσουμε να τα δαπανίσουμε για το περιβάλλον τα λοιπά, γιατί θα πέφτουν στη διπλή ενίσχυση. Γιατί αν το έχουμε ως στόχο στον πρώτο πυλώνα, τότε δεν μπορώ να το μεταφέρω στο δεύτερο πυλώνα. Έχουμε μεγάλη ανάγκη για συζήτηση ακόμα, αλλά η αντιπρόεδρος, η κυρία Μακίνες, δυστυχώς δεν μπορεί να είναι παρούσα και ζητεί συγγνώμη, γιατί στο Δουβλίνο ε, συμμετέχει στην απονομή ενός ε, βραβείου όπου τιμάται ο πρώην ε, Πρωθυπουργός σας, ο κύριος Κένι. Και μου είπε να σας ρωτήσω το εξής. Η πρότασή σας είναι αρκετά ισχυρή έτσι ώστε να αντέξει τις επιπτώσεις του Brexit στις γεωργικές αγορές. Εγώ θα έχω αρκετό χρόνο για να σας κάνω τις ερωτήσεις μου κύριε Επίτροπη στη συνέχεια. Επόμενος συντονιστής. Ευχαριστώ κύριε Επιτροπέ, ο κύριος Αντρίου. Όχι, δεν είναι ούτε φιλόδοξη, ούτε ισορροπημένη η πρότασή σας, ούτε καν ρεαλιστική. Και βεβαίως δεν λαμβάνει υπόψη τις μεταλλάξεις που συμβαίνουν στον κόσμο. Είπατε λιγότερο από 12% σε πραγματικές τιμές. Εμείς προχωρούμε, αλλά λέτε λιγότερα για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Δεν ξέρω, μήπως μας δώσετε κάποια στοιχεία παραπάνω. Όχι, κύριε Επίτροπε. Ε, είναι το πιο ευέλικτο πλαίσιο για τα κράτη-μέλη για να έχετε μια σύντομη συμφωνία το συντομότερο δυνατόν. Ωστόσο, δεν μας λέτε τίποτα για την ουσία από την αρχή της δεκαετίας του 90. Τι βλέπουμε, σύνδεση, απαγκίστρωση ε, των ε, ενισχύσεων και ευθυγράμμιση στις διεθνείς τιμές, η στρατηγική ε, του ελάχιστου κοινού παρονομαστή. Νομίζω στη συνθήκη της Λισαβόνας χρειάστηκε για να έχει λόγο το Κοινοβούλιο στα γεωργικά. Και τώρα αποφασίζετε να μας βγάλετε ε, off-site γιατί το Κοινοβούλιο δεν έχει κανένα λόγο όταν πρόκειται για κρατικές ε, ε, ε, πολιτικές. Πρόκειται λοιπόν για τη διαχείριση κρίσεων και εκεί ακριβώς είναι το πρόβλημα. Η φιλελεύθερη πολιτική μπορεί να είναι θεμητή, αλλά δεν αρκεί για να αποζημιώνει τους αγρότες και να τους ανταμείβει. Και σε περίπτωση κρίσης αγοράς θα πρέπει να ε, επεμβαίνεται. Αυτό θα πρέπει να γίνει μόνο σε κοινοτικό επίπεδο, η διαφύλαξη της εσωτερικής αγοράς. Δυστυχώς βλέπουμε επανεθνικοποίηση και εγώ έτσι εξακολουθώ να την αποκαλώ. Επανεθνικοποίηση της κοινή γεωργικής πολιτικής. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε δεν θα ε, ε, αναλωθώ σε ευχαριστήσεις, θα πάω κατευθείαν στο ψητό. Η Γεωργία, όπως τη γνωρίζουμε, είναι ένας κλάδος της οικονομίας που όταν θεωρεί κανείς ότι όλα πάνε καλά, ξαφνικά κάτι συμβαίνει ε, που το δημιουργεί, προκαλεί πολλά προβλήματα του αγρότη χωρίς να φταίει καθόλου εκείνος. Τα τελευταία χρόνια έχουν συμβεί πολλά δεν μπορούμε να καθίσουμε λοιπόν και να αγγίθουμε τι θα κάνει η επόμενη γεωργική πολιτική. Θα πρέπει να έχουν ευελιξία αγρότε και εργαλεία για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τι προκλήσει που του περιμένουν. Και θα ήθελα να μάθω περισσότερα για το πώ προτίθεστε να ζητάτε διευκρινήσεις από τα κράτη-μέλη λέει ο κύριος Νίκολσον, ε, για ε, αυτό το σώμα το ενιαίο συντονιστικό και συνεργασία πώς θα γίνεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί φοβούμε ότι τώρα αυτό που φτιάχνουμε άλλο ένα τέρας γραφειοκρατίας και οι αγρότες θα πληρώσουν τα σπασμένα και θα πρέπει να δικαιολογούνται για την κάθε τους ενέργεια. Και ποια σχέση θα έχει αυτό ε, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με το κράτος μέλος και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ξέρω ότι πολλά από αυτά τα πράγματα θα διευκρινιστούν σε επόμενους μήνες. Κάνατε ένα σχόλιο προηγουμένως για το τελικό αποτέλεσμα θα πρέπει να είναι υπέρ του αγρότη. Με περί αυτού πρόκειται. Εγώ έχω δει μεταρρυθμίσεις από το Μαξάρι, τον Φίσλερ, Φίσερ Μπόλ και τώρα τη δική σας. <laughs> πραγματικά πολλοί κόσμος. Αλλά όταν συζητάμε για τον προπολογισμό, ορισμένοι λησμονούν το εξή. Όταν μεταρρυθμίστηκε η κοινή γεωργική πολιτική για τις πολιτικές, ε, δεν είχε καμία αριθμική προσαρμογή ούτε σύνδεση με τον πληθωρισμό. Δηλαδή κάθε χρόνο σε πραγματικές τιμές χάνουν λεφτά οι αγρότες και αυτό τσιμωδιά. Και πρέπει να σας πω, τα χρήματα αυτά τα έχουν βγάλει ή αγελαδοτρόφοι ή ε, πρόβατο τρόφι και λυπή κτηνοτρόφι. Και εγώ δεν θέλω να δω να χάνονται ε, οι, γαλακτο, ε, ε, οι αγελάδες και η γαλακτοπαραγωγή από τα, τις business που κάνετε και τις συμφωνίες με το Μεκροσού. Μερκοσού. Ο πρόεδρος. Μιλάτε για φιλελευθερισμό, αλλά αυτός ο φιλελευθερισμός δεν είναι η τελευταία μεταρρύθμιση, είναι επί περίοδου Fisher Ball. Σε αυτό ανάγεται. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε για τα όσα μας είπατε και τα όσα μας προσφέρατε. Να παραμείνετε σε επαφή μαζί μας και να συζητήσουμε αν έχετε ή αν έχουμε εμεί ερωτήσεις. Για μένα είναι πολύ σημαντικός ο προϋπολογισμός για να καταλάβουμε τι θα γίνει αν δεν προλάβουμε γέρο και δεν έχουμε τον προϋπολογισμό. Θα υπάρξει κάποια μεταβατική περίοδος ή μήπως θα πρέπει οι αγρότες ε, στο μέλλον να περιμένουν περικοπές αν δεν έχει ολοκληρωθεί και προταθεί ο προϋπολογισμός. Μιλήσατε και για στρατηγικά σχέδια. Ακούω ότι θα υπάρξει μια ομάδα δράσης task force που θα υποστηρίζει τα κράτη-μέλη. Πραγματικά επιγόντως μας χρειάζεται μια τέτοια ομάδα. Ε, θα προτείνετε όμως συγκεκριμένα μέτρα για το πώς όλα αυτά θα εφαρμοστούν στην πράξη. Και θα μας ενημερώσετε για τα στρατηγικά αυτά σχέδια. Επιπλέον, ε, ε, μιλήσατε για την απλούστευση, αλλά ε, ζητάτε ετήσια σχέδια και ε, απολογισμούς από τις κυβερνήσεις. Πού τη βλέπετε την απλούστευση αυτή για τους αγρότες τελικά και για την ρεσιμότητα. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι ακόμα. Ε, έχετε συμπεριλάβει εκεί ε, και την παροχή συμβουλών και την υποστήριξη από τα κράτη-μέλη, γιατί σε πολλά κράτη-μέλη δεν έχουμε συμβουλέ. Και για το κάπινγκ, αυτή την ε, ανώτατη, την οροφή, ε, και αυτό μας προβληματίζει. Πώς θα αποτρέψετε στο μέλλον να σπάει μια επιχείρηση αγροτική. Όλα αυτά μας ταλαιπωρούν και μας προβληματίζουν. Γενικά, δεν τη βλέπω τόσο αρνητικά αυτή την εξαγγελία σας. Υπάρχουν και ευκαιρίες που θα πρέπει να τις αξιοποιήσουμε και να συνεργαστούμε όλοι προς την κατεύθυνση αυτή για να προκύψει κάτι καλό για τους αγρότες και για τις μικρομεσαίες γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Ευχαριστώ. Κάθε επίτροπος της κοινή αγροτικής πολιτικής συγκρίνεται σε σχέση με τον ε, προηγούμενη μεταρρύθμιση. Έχουμε ε, λιγότερους νεαρούς αγρότες ε, και φυσικά ακούμε πολύ συχνά εδώ τον αριθμό ότι το 80% των ενισχύσεων πάνε στο 20% των πιο πλούσιων αγροτών. Και γνωρίζουμε όλοι ότι ο μόνος τρόπος που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε παρκώς αυτή την ανισότητα είναι να βάλουμε ένα ανώτατο όριο στις ενισχύσεις που μπορούν να ληφθούν. Και όλοι ε, είδαμε τα έγγραφα που έλεγαν ότι η Κομισιόν επιτέλους θα πρότεινε ένα ανώτατο όριο 60.000 στις πληρωμές. Δυστυχώς η πρότασή σας όταν δημοσιεύτηκε είναι γεμάτη κενά και ε, οποιαδήποτε επίπτωση των πληρωμών είναι οφθαλμαπάτη. Είπατε ότι θέλετε να δώσετε προτεραιότητα στην, ε, στις άμεσες πληρωμές. Εγώ θα έλεγα ότι και πάλι ουσιαστικά δίνεται προτεραιότητα ε, στους, ε, στα συμφέροντα των μεγάλων αγροτών. Επίσης για τους νέους αγρότες αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί θέλουμε ένα μέλλον για την Ευρωπαϊκή Γεωργία και πάλι οι άνθρωποι αυτοί βρίσκονται ε, στο έλεος ε, του αποθεματικού γιατί ε, εξακολουθεί να παραμένει ένα σύστημα δικαιωμάτων σε ισχύ. Ο όρος ε, απλούστευση δεν αναφέρθηκε στην Επιτροπή. Αν ε, θέλουμε να απλουστεύσουμε τις πληρωμές, έχουμε έναν ορισμό ε, για τον ενεργό γεωργό, για την επιλέξιμη γη. Γιατί να μην αναφέρουμε και τα μέτρα όπου θα έχουμε front loading σε πληρωμή ανακτάριο. Ξέρετε, ε, η μεγάλη πλειοψηφία των γεωργών με κάτι τέτοιο θα ήταν σε πολύ καλύτερη θέση και οι αγροτικές κοινότητες ε, θα λάμβαναν ε, πολλά οικονομικά κίνητρα και οι μόνοι που θα μπορούσαν να φέρουν αντίρρηση σε αυτό ήταν αυτοί που έχουν πολύ μεγάλα συμφέροντα εταιρικά και ουσιαστικά απομιζούν το σύστημα της κοινή γεωργικής πολιτικής. Κύριε Επίτροπε, συγχαρητήρια. Ωραία τα λόγια. Αλλά η πολιτική είναι ίδια παλιά με νέο περιτύλιγμα και το περιβάλλον υποφέρει από αυτή την κοινή γεωργική πολιτική. Χάνουμε εκατοντάδες χιλιάδε αγρότες, οι εργαζόμενοι στη γεωργία δεν έχει διερμηνία. Έχει. Ε, υποφέρουν από αυτή την πολιτική και το αποτέλεσμα είναι μία από τα ίδια. 80% των πληρωμών πηγαίνουν στον πρώτο πυλώνα και τα πάντα παραμένουν όσοι είχαν. Μιλάτε για την κατάργηση του πρασινίσματος και ε, ε, για φιλόδοξα νέα περιβαλλοντικά μέτρα. Ποια είναι αυτά και πώς θα διαμορφωθούν. Πιστεύετε σοβαρά ότι θα φροντίσουν τα σχέδια των κρατών μελών να γίνει μια φιλόδοξη περιβαλλοντική πολιτική και στην ε, περασμένη μεταρρυθμίση βελτιώσαμε. Μάλλον αποδυναμώσαμε το πρασίνισμα και τώρα το καταργούμε τελείως. Δεν τα πιστεύετε το ίδιο αυτά που μας λέτε. Και επίσης μπορείτε να μας εξηγήσετε πώς αυτές όλες οι συμφωνίες που θέλετε να κάνετε ε, συνάδουν με την πολιτική μας. Δεν μπορούμε να ανοίξουμε όλες τις αγορές στην Ευρώπη για πιο φθηνή παραγωγή. Δεν βγαίνουν αυτές οι εξισώσεις και για την περιβαλλοντική πολιτική. Πραγματικά ε, έχω ξοργιστεί για τις περικοπές στο δεύτερο πυλώνα. Ας είστε ειλικρινείς και πείτε ε, πραγματικά στοιχεία 25% όχι 15%. Είδηση δεν θα πάρουν ε, οι κυβερνήσεις και θα καταστρέψουμε όλα τα περιβαλλοντικά. Μιλάτε για ανώτατα όρια. Ξέρετε ότι υπάρχουν πέντε μεγάλες χώρες που θα αρνηθούν και αυτά είναι σχέτη ρητορική. Λοιπόν, το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι αμέσω να αποσύρετε την πρότασή σας και να φέρετε καινούρια ε, και να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας από μια πολιτική που έχει αποτύχει και να μην συνεχίσουμε τύχες Γιάννη τύχα πάντα. Στο τέλος δεν θα μας πιστεύει η ψυχή αν συνεχίσουμε σε αυτό το δρόμο. Να μας ξανάρθετε σε λίγες εβδομάδε και να μα φέρετε τίποτα καινούργιο, αυτό θα ήταν το καλύτερο. Βλέπω ότι... Βλέπω ότι άλλαξε λίγο η διάθεσή σας. Προσέξτε. Εμένα με ενδιαφέρει η πρόταση αυτή σε ό,τι αφορά το κλίμα. Ποιο... Ε, εδώ θα συμπεριληφθούν οι ατμοί του νερού, πόση η μείωση των αερίων θα μετρηθεί Πώς γνωρίζουμε ότι αν έχουν γίνει μειώσεις σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Το ίδιο ισχύει και για τις εκπομπές ότου. Εδώ έχουμε μια αντίφαση. Ο Επίτροπος θέλει μια αύξηση των καλλιεργειών, εδώ έχουμε μια αύξηση των εκπομπών. Πώς θα μετρηθούν όλα αυτά. Και αν υποθέσουμε ότι υπάρχει μία επιδείνωση, σε τι βαθμό θα οφείλονται οι εκπομπές των θερμοκηπίων που θα ε, αποδοθούν ε, στην, στον, στον ουρανό, στον ε, ήλιο, στο φεγγάρι. Συνεπώς, πραγματικά χρειαζόμαστε ένα χρήση οδηγίας για το πώς θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε το καιρό. Ενδεχομένω, οι αγρότε θα παρανομήσουν, γιατί πραγματικά δεν υπάρχει τρόπο συμμόρφωση σε αυτά που ζητάτε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σοζόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πιστεύω ότι η γεωργία θα πρέπει να βρίσκεται στην καρδιά της ΚΑΠΑ θα πρέπει να μας απασχολήσει το μέλλον της ε, ΚΑΠΑ στο μέλλον. Στην ε, Γαλλία λέμε τα πράγματα κατερεύσουν σε 10 χρόνια. Θα ήθελα να πιστήσω την προσοχή σας στην ε, δυνατότητα μεταφοράς κονδυλίων από τον ένα πυλώνα στον άλλον. Η Επιτροπή θέλει μία πολιτική περιβαλλοντική ή μία πολιτική γεωργική Ξέρετε ότι μιλώντας για τις επιδόσεις των περιβάλλον στο άρθρο 123 θα μπορούσαμε να εγγυηθούμε ότι αυτό θα έχει επίπτωση στα έσοδα των γεωργών, στο εισόδημα των γεωργών, πολύ το αμφιβάλλω. Σε ό,τι αφορά την απλοποίηση της ΚΑΠΑ, πραγματικά δεν, δεν το πιστεύω. Πιστεύω ότι θα υπάρχει όλο και μεγαλύτερη γραφειοκρατία. Ε, τώρα μιλάμε για το άρθρο 68. Η κοινωνική πολιτική ήταν θέμα των κρατών μελών και παρόλο το ΣΕΝΚΕ, παρόλες τις αυταπάτες που υπήρξαν, υπάρχουν ορισμένα πράγματα κυριαρχίας που δεν μπορούν να ξεπεραστούν. Στην ουσία ήταν από τα κράτη να αγοράσουν τις γεωργικές γέες. Δεν μπορούμε να επενδύσουμε στη γη μας όταν επιτρέπεται η κερδοσκοπική επένδυση από holding που δεν έχουν κανένα απολύτως ενδιαφέρον για τους γεωργούς. Κύριε ε, Επίτροπε, σας εγγυώμαι ότι τα τρία αυτά σημεία που έδειξα δεν είναι τα μοναδικά που μας απασχολούν. Ευχαριστώ. Κυρίε και κύριοι, όπως σας είπα, θα δώσω το λόγο και πάλι στον Επίτροπο για τις απαντήσεις. Ευχαριστώ. Καταρχήν ε, για το νέο ε, μοντέλο υλοποίηση ε, που έχει να κάνει με το πώς το σχεδίσαν οι Κομισιόν και τα κράτη-μέλη στην σημερινή πολιτική που συμφωνήθηκε το 2013 υπάρχει σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Γιώργου και όλα τα κριτήρια και οι κανόνες επιλεξιμότητας για οκτώ προγράμματα που εφασίζονται από την Ευρώπη και υπάρχει μια προσέγγιση ε, κοινή διαχείριση μεταξύ Ένωση και Μελών για την εφαρμογή. Τώρα, αυτό που ζητάμε με τα σχέδια στρατηγικά σχέδια της ΚΑΠ. Τα κράτη-μέλη είναι ότι θα παρουσιάσουν επαρκή ευελιξία για να μπορέσουν να προσαρμοστούν στις δικές τους τοπικές συνθήκες. Πώς θα μπορέσουν να πετύχουν τους ε, νέα κύριους στόχους της ΚΑΠ που θα πρέπει να εγκριθούν από ολόκληρο το Σώμα των Επιτρόπων, όχι μόνο από τον Επίτροπο Γεωργίας, σε σχέση δηλαδή με το αν ε, γίνονται σεβαστές οι υποχρεώσεις που τίθενται στα κριτήρια. Αυτή είναι η θεμελιώδης λέγει ότι η Ευρώπη ε, δεν ε, θα ε, αποφασίζεται κάθε λεπτομέρεια, αλλά αυτά θα αποφασίζονται στα κράτη-μέλη και επίσης και στόχοι θα τίθενται σε επίπεδο κράτους μέλους. Θέλω να το τονίσω αυτό. Επομένω, δεν ξέρω πώ θα υπάρχει μεγαλύτερη γραφειοκρατία, γιατί οι περισσότεροι κανόνε που έχουμε σήμερα, που ουσιαστικά επικαλύπτονται με κανόνε κρατών μελών, έρονται. Έτσι λοιπόν, υπάρχει μια μεγάλη διαφορά, μια μεγάλη αλλαγή σε σχέση με την μείωση των κανόνων που πρέπει να σεβαστούν οι γεωργοί. Για πρώτη φορά, και το κύριο Ντέ, οι νεαροί αγρότε ε, είναι ένα από τα εννιά κριτήρια, ένα από του εννιά στόχου για την ανανέωση τη γενιά. Έτσι λοιπόν, αν κάνουν ήδη κάποια καλή δουλειά τα κράτη-μέλη, το χάρη στολίζουν εταιρικέ σχέσει, στη φορολογία, αυτό θα ληφθεί υπόψη στη στρατηγική που πρέπει να εκπονήσουν και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δώσει πρόσθετη αξία, ε, προσθέμενη αξία στα κρατη έχουν τουλάχιστον ένα καλό σχέδιο για το πώς μπορούν να έχουν καλύτερα αποτελέσματα για τους νέους γεωργούς. Έχουμε μόνο 6% γεωργούς κάτω των 35 ετών που ελέγχουν τις εκμεταλλεύσεις. Αυτό είναι λοιπόν ένα σημαντικό στοιχείο. Στην έκθεση Dortman ε, έχουμε 197 προτάσεις. Συγγνώμη, 187 175 μας βρίσκουν σύμφωνος επί της, αρχές, επί της αρχής. Οι άλλες 12 έχουν να κάνουν με τα χρήματα. Φυσικά τα χρήματα είναι πολύ σημαντικά για τους αγρότες, αλλά σε σχέση με το τι μπορούμε να προτείνουμε, αυτό μπορούμε να κάνουμε καλύτερο αρχικά. Και φυσικά τώρα είναι ανοιχτό για τη συζήτηση για το πολιτικό δημοσιονομικό πλαίσιο για να προσπαθήσουμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Αλλά δεν είναι κακό αποτέλεσμα 175 στις 187 όταν ξεκινά αυτή η Επιτροπή της Εργασίας σας. Ε, κύριε Άντριου, διάβασα και το έγγραφο που μου δώσατε από τους σοσιαλιστές ε, πολύ προσεκτικά και η απορρίθμιση στην οποία αναφερθήκατε ήδη είναι ε, μέρος της νομοθεσίας που εγκρίθηκε την περασμένη φορά, το χάρη, προσανατολισμό στην αγορά. Αν ε, το αλλάξετε αυτό, πρέπει να καταθέσετε ουσιαστικέ τροπολογίε. Όμω, ε, θα πρέπει να έχουμε κάποιο τρόπο να παρέμβουμε. Συμφωνώ μαζί σα και αυτό αναφέρεται ρητά στο εγγραφό σα. Γι' αυτό το καθιστούμε υποχρεωτικό να υπάρχουν εργαλεία διαχείρισης κινδύνου που θα βασίζονται στο Omnibus. Αυτό είναι μεγάλη βελτίωση για να βασιστούν στην διαπραγματευτική δύναμη ε, του Γεωργού και στην νομοθεσία για τους θεμητούς ε, κανόνες και να βασιστούν στην ε, διαφάνεια της αγοράς που θα έχουμε αργότερα. Έτσι λοιπόν υπάρχουν όλες οι προτάσεις για τη διαχείριση. Τη κρίση. Υπάρχουν και τα εργαλεία διαχείριση κρίση και πρώτη φορά καθίστανται υποχρεωτικά και όλα όσα σας ανησυχούν υπάρχουν στην πρόταση. Κυρία Νίκολσον, ε, αναφέρθηκα νομίζω στην ερώτησή σας ότι είναι μια αλλαγή σε μια προσέγγιση που θα βασίζεται στους γεωργούς ε, θα έχουμε ε, ουσιαστικά άμεση δραστηριότητα των εργών και αυτή τη στιγμή έχουμε πολλά κρατημέλη έχετε δίκιο. Πρέπει να δούμε το θέμα του κανονιστικού υπερθεματισμού. Εσείς ε, ξέρετε ότι ποτέ δεν υπήρχε τη αριθμική προσαρμογή ε, των πληρωμών. Αυτό είναι ένα θέμα της Επιτροπής Προπολογισμού και δικό σας θέμα να το επιλύσετε. Όμως ε, έχουμε τις τρέχουσες τιμές, παραδείγματος χάρη. Αν εγώ πληρώνω 500 ευρώ το μήνα για 20 χρόνια, είναι η ίδια αρχή που υπάρχει στο επιταστές πρόγραμμα για την ΚΑΠ. Αυτές είναι οι τρέχουσες τιμές ε, και αυτό θα είναι ο έλεγχος ε, που θα γίνει το 2021 σε σύγκριση με το 2020 και τρέχουσες και σταθερές τιμές ε, δεν έχει σημασία για τους γεωργού. Θέλουν τελικά να δουν τι παίρνουν. Όμως φυσικά καλωσορίζουμε περισσότερα χρήματα από οπουδήποτε. Είναι πάρα πολύ ρομαντικό να μιλάει κανεί για χρήματα. Πολύ ωραία, Πρόεδρε. Υπάρχει και μια διάταξη, μια πρόβλεψη στην πρόταση για μια πιο τομεακή προσέγγιση για να αντιμετωπίσουμε τα θέματα για τον τομέα ε, του βοηοκρέατος και ποιον άλλο τομέα. Υπάρχει σήμερα ε, ουσιαστικά μια πρόταση να δούμε, να, τα, να υιοθετήσουμε μια πιο τομεακή προσέγγιση. Γιατί υπάρχουν πολλοί τομείς που δέχονται πίεση αναφάσεις. Φυσικά τα κονδύλια είναι πολύ σημαντικά και θα πρέπει να δώσουμε βεβαιότητα στους Γιώργους μας. Είμαστε σε επικίνδυνους ε, καιρούς λόγω του Brexit. Ε, στα τέλη ε, Μαρτίου μπορεί να έχουμε κατάρρευση των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Βρετανία. Τι θα κάνουμε για να διασφαλίσουμε τη χρηματοδότηση των, προγραμμάτων μα. Θα πρέπει να το σκεφτούμε πολύ σοβαρά και ξέρω αυτό κάνει η Επιτροπή Προπολογισμού αυτή τη στιγμή και θα πρέπει να συνεργαστούμε μαζί του για να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει συνέχεια των πληρωμών. Και πώς ε, τελικά θα καλύψουμε αυτό το κενό των 12 ε, εκατομμυρίων. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτό το θέμα και να υπάρξουν και κάποιε συμβουλέ. Ε, να δεχτούμε κάποιες συμβουλές. Αυτό κάνω αυτή τη στιγμή. Εμείς θα δώσουμε πολύ περισσότερες ε, πληροφορίες για τα στρατηγικά σχέδια. Τώρα, για τις επιδόσεις. Ρωτήσατε για τις επιδόσεις και πώς θα λειτουργήσει αυτό το θέμα. Έχουμε αιτήσιες εκθέσεις αυτή τη στιγμή από τα κράτη-μέλη σε σχέση με τις επιδόσεις. Έχουμε 200 δείκτες αυτή τη στιγμή. Ζητάμε πληροφορίες από τα κράτη-μέλη για αυτούς τους δείκτες και φυσικά αυτά θα πρέπει να εξορθολογιστούν και να μειωθούν και ουσιαστικά να υπάρχει ε, κάποιο νόημα για το Γιώργο ως προς τις ε, επιδόσεις. Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να δείξει ότι έχει συμβουλευτικές υπηρεσίες. Και σε σχέση με το ανώτατο όριο, φυσικά αυτό είναι ένα μεγαλύτερο θέμα για κάποια κράτη-μέλη, υπάρχουν διατάξεις στον για το πώς θα εφαρμοστεί αυτό. Ε, τώρα εξαρτάται από τα κράτη-μέλη, αν θα θέλουν να έχουν 60.000. Ε, τώρα έχουμε 150.000 ακούσια βάση σε πολλά κράτη-μέλη. λοιπόν το θέμα είναι αν θέλετε υποχρεωτικό ή ακούσιο. Όμω εγώ είμαι υπέρ τη ε, ισότιμη κατανομή των πληρωμών και έχω προσπαθήσει να το κατοπτρίσω αυτό. Ε, τώρα η αρχή είναι ένα θέμα για τα κράτη-μέλη αν θέλουν να συνεχιστούν τα δικαιώματα ή όχι. Ε, μπορεί να τιμωρηθούν αν επιθυμούν να συνεχίσουν κάτι τέτοιο ε, και ίσως να πρέπει να αλλάξουν ε, σε ένα νέο σύστημα. Τώρα υπάρχει το σύστημα στραματικών ενισχύσεων. Ίσως Μπορεί να θέλετε να είστε στην κυβέρνηση σύντομα και μπορείτε να επιμείνετε ε, με οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα ή σε συνασπισμό βρεθείτε. Οι νεαροί γεωργοί, όπως ανέφερα νωρίτερα για πρώτη φορά, θα αποτελούν τμήμα ενός συγκεκριμένου στόχου. Τα κράτη-μέλη έχουν πείσει την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι κάνουν κάτι αληθινό. Έχουμε κάποια μέτρα απλούστευσης. 5.000 ε, αγρότες στην Ιρλανδία εποφελήθηκαν πέρσι από τον έλεγχο προ-πρόληψης, δηλαδή ήταν ένα μέτρο αυτό, φυσικά πρέπει να κάνουμε παραπάνω. Και αυτή είναι μια θεμελιώδες ε, αλλαγή στην εφαρμογή της πολιτικής, γιατί θέλαμε κανονιστικό υπερθεματισμό από τα κράτη-μέλη. Έχουμε λοιπόν μια ευκαιρία όταν παρουσιάζονται τα σχέδια να μπορούμε να τα εξετάσουμε λεπτομερώς ε, και φυσικά να υπάρχουν πλουστεύσεις όχι μόνο για την Κομισιόν και τη Δίκηση αλλά και για τους αγρότες. Κύριε Χόσλινγκ, δεν ε, διαφάσετε τα έγγραφα πριν έρθετε στη συνεδρίαση γιατί θα δείτε ότι περιγράφεται εκεί η αρχιτεκτονική πρασινίσματος. Τώρα πρέπει να σας ε, τα εξηγήσω όλα εγώ. Διαβάστε τα έγγραφα σας παρακαλώ. Η νέα αρχιτεκτονική της ΚΑΠ είναι αρκετά φιλόδοξη. 20% ε, mainstream είναι αυτή τη στιγμή οι κλιματικές ε, δράσεις. Ε, είναι κάτι πολύ καλό για το μέλλον. Η έκθεση που έχουμε από το ελεκτικό συνέδριο για το πρασίνισμα δεν, μας λέει ότι δεν έχει λειτουργήσει. Έτσι λοιπόν τώρα δίνουμε μια προσέγγιση με κίνητρα για τα οικολογικά ε, καθεστώτα στον πυλώνα 1 και πολύ συχνά το έχετε ζητήσει, τώρα το κάνουμε. Και κατόπιν η φιλοδοξία. Αν θέλουν οι άνθρωποι να πάρουν περισσότερα χρήματα στον πυλώνα 2, πρέπει να εφαρμόσουν ε, περιβαλλοντικά μέτρα. Έτσι λοιπόν ε, δεν ε, παρουσιάζω νέες προτάσεις. Ε, εσείς να παρουσιάσετε τις τροπολογίες σας και θα τις εξετάσουμε που θα κάνουμε και με τις άλλες πολιτικές ομάδες. Κύριε Άγνιου, η κυρία Αλλαγή έχει να κάνει με τα κράτη-μέλη παρά με το Γιώργο. Υπάρχει πολύ φυσταμένη νομοθεσία που αναφέρεται που θα πρέπει ήδη να εφαρμόζεται από τα κράτη-μέλη. Ένα καλό παράδειγμα είναι τι έγινε στις κάτω χώρες, όπου η φυστάμενη νομοθεσία ε, ουσιαστικά εφαρμόσε ε, μέτρα για το γαλακτοκομικό τομέα ε, και έπρεπε ουσιαστικά να μετρήσουν 160.000 αγελάδες σε κάτω χώρες, σφάξουν 160.000 αγελάδες, με συγχωρείτε. Και φυσικά δεν ε, ήταν κάτι επιθυμητό, δεν τους άρεσε. Θα σας ε, ενημερώσει ο κύριος Χόσλινγκ για okay. τις λεπτομέρειες. Ο κύριος Χότιμα θα σας ενημερώσει για τις εξελίξεις. Η πολιτική, κύριε Χουαζού, είναι οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντική. Υπάρχουν τρεις κύριοι στόχοι που πρέπει να γίνονται σεβαστοί. Και θα πρέπει να καταβάλουν την ισχύ στους γεωργούς για όλους αυτούς και φυσικά θα πρέπει να υποστηρίζουμε τις αγροτικές κοινότητες ως και ως προς τις υποδομές. Εγώ θα ήμουν ικανοποιημένος να υπήρχαν περισσότερα κονδύλια για την ΚΑΠ και εξήγησα το πλαίσιο στο οποίο βασίστηκε αυτή η σημερινή πρόταση. Όμως είναι μια αρχική θέση, είναι μια διαπραγμάτευση και τα κράτη-μέλη ε, λένε ότι δεν θέλουν να έχουν πλέον κόστος ε, και το καλωσορίζω. Ελπίζω να υπήρχε ομοφωνία από τα κρατη Θα δούμε. Αυτά προς το παρόν. Ο πρόεδρος, ε, ωραία. Τώρα δεύτερος γύρος, έχω να κάνω δύο σχόλια. Όταν δίνουμε κάποιες αρμοδιότητες ε, σε κάποιες χώρες, δεν σημαίνει ότι καταργούμε την κοινή γεωργική πολιτική. Απλώς παίρνει κάποιες αρμοδιότητες η χώρα. Δεν είναι αυτό. Το δεύτερο, για τους νέους αγρότες. Τα κράτη-μέλη παίζουν και εκεί ένα σημαντικό ρόλο ε, για το πώς μεταβιβάζονται οι αγροτικές γιές, για το πώς φορολογούνται οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Ε, αυτά είναι θέματα που πρέπει να τα δούμε ευρύτερα. Να δώσω και μια απάντηση. Ο κύριος Μάτο, ευχαριστώ πολύ. Ε, στα Κανάρια, κύριε Επιτροπέ, ανησυχούμε βαθύτατα. Ο πρόεδρος Γιούνκερ πριν από λίγους μήνες ε, στον αντίστοι, στην αντίστοιχη σύνοδο στη Γουιάννα είπε θα συνεχίσουμε τα προγράμματα ΠΟΣΕΙ και δεν σκεφτόμαστε ούτε να τα μειώσουμε ούτε να τα διορθώσουμε προς τα κάτω. Και στο Κοινοβούλιο πριν από λίγο καιρό, τον περασμένο μήνα, εγκρίναμε ένα ψήφισμα που ζητούσαμε αύξηση του προπολογισμού ΠΟΣΕΙ για την περίοδο 2021-2027. Απέναντι σε αυτό, ποια είναι η πραγματικότητα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε να μειωθεί κατά 3,9% ετησίω η πρικοδότηση ΠΟΣΕΙ. Αν αυτό επιβεβαιωθεί, που ελπίζω να διαψευστεί, θα έχει δραματικές συνέπειες για τη γεωργία μας, για το περιβάλλον μας, για τη γεωργία μας. Και από πάνω ε, είναι κατάφορη ε, παραβίαση του άρθρου 349 της συνθήκης. Επίσης, να μειωθούν ε, τα μέτρα τα αντισταθμιστικά για την ανάπτυξη της υπαίθρου που ήταν 85% και τα πάτε στο 70%. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Κύριε Επίτροπε, σας παρακαλώ να δεσμευτείτε ότι ε, ε, θα τηρήσετε το λόγο του κυρίου Γιούγκερ. Μπορεί να φαίνεται ότι 25 εκατομμύρια ευρώ δεν είναι και πολλά λεφτά για την ε, ΚΑΠ και το σύνολό της, αλλά για τις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες είναι θέμα επιβίωσης αυτό. Είναι το πάνε. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σε ένα λεπτό θα ήθελα να εκφράσω δύο σκέψεις. Η πρώτη αφορά τον προπολογισμό και θα ήθελα να εκμεταλλευτάω την παρουσία του πρόεδρου του Υπάρχουν έξι υπουργοί γεωργία οι οποίοι υιοθέτησαν μια θέση προσπίζοντα τον προπολογισμό της ε, κοινή αγροτική πολιτικής. Ελπίζω ότι ο αριθμό αυτό θα αυξηθεί στο επόμενο Γεωργικό Συμβούλιο εμείς ως Επιτροπή, ως Κοινοβούλιο θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι στηρίζοντας αυτή την πρωτοβουλία έτσι ώστε να μπορέσουμε να αποσπάσουμε καλύτερες συνθήκες γιατί όπως είπαμε πολλές φορές αυτή την Επιτροπή δεν είναι σωστό για τους γεωργούς ε, να πληρώνουν την ε, απόλυτα θεμητή επιλογή των Βρετανών σε ό,τι αφορά την ΚΑΠΑ, θα ήθελα να θυμίσω ότι δεν τίθενται υποσυζήτηση οι θετικές ειδήσει που μας μετέφερε ο Επίτροπος. Η ελαστικότητα μας αρέσει, το θέμα των μικρών γεωργών μας αρέσει, η ενδυνάμωση ε, των διαχειριστικών εργαλείων μας αρέσει. Το θέμα είναι η εγκατάσταση. Έχουμε την εντύπωση ότι ε, η όλη δομή Δηλαδή ότι θα δημιουργηθεί περισσότερη γραφειοκρατία και περισσότερες δυσκολίες, ιδιαίτερα σε χώρε σαν τη δική μου που πλήττονται από την γραφειογραφία. Ευχαριστώ, ευχαριστώ όλους και τον Επίτροπο. Συμφωνώ με όσα υπόθηκαν από τον κύριο Δεκάστρο και όσα είπε ο συνάδελφος Ντες γιατί πιστεύω ότι με αυτή την πρόταση ε, πέρα πολύ μακριά από τη μείωση του διοικητικού άχθους ε, ουσιαστικά ε, τι κάνουμε, αυξάνουμε την γραφειοκρατία αλλά δημιουργούμε και ανασφάλεια δικαίου. Επίσης πιστεύω το εξή. Μα είπε ο Επίτροπο ότι θα πρέπει να προσανατολιστούμε προ την αγορά με τα κατάλληλα εργαλεία διόρθωση. Εμένα θα μου άρεσε να υιοθετηθεί αυτή η πρόταση που έχουμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον τομέα των εγωπροβάτων ε, και ε, είχαμε κάνει κάποιο αίτημα σε μια έκθεση πρωτοβουλία. Επίση, θα ήθελα να μου πείτε τι γίνεται και με την κτηνοτροφία στα νησιά. Υπάρχουν πάρα πολλέ δυσκολίε και δεν είναι άκρο από μα περιοχέ, όμω έχουν πάρα πολλά μειονεκτήματα. Και θα ήθελα να δω και κάτι παραπάνω για του νέου γιατί δεν έχουμε καμία καινοτομία να τους προσφέρουμε πέρα από το τι μπορούμε να φανταστούμε σε αυτό το νοικό. Έχουμε λοιπόν μια μεγάλη πρόκληση, κυρία Χόιμπους. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πίτροπε, τώρα επανειλημμένα μας είπατε ότι δεν θα υπάρξει επανεθνικοποίηση της ΚΑΠ, αλλά έχετε ορίσει κάποιους κοινούς στόχους που πάνω κάτω θα ισχύουν το ίδιο για όλους. Αν κοιτάξω αυτούς τους στόχους όμως είναι πάρα πολύ διαφορετικοί για να μην πω και αντιφατικοί εν μέρη. Και αν έρθουν τώρα τα κράτη να διαλέγουν εκείνο που τους αρέσει, που είναι πιο ανταγωνιστικό και τα λοιπά, είναι καλύτερο το προτιμώ από το περιβάλλον ή από το κλίμα, τότε θα μπούμε σε μια κατρακύλα. Ακόμα και οι δείκτες τους οποίους ορίζεται είναι πάρα πολύ αδύναμοι και δεν έχουμε σαφή εικόνα. Δηλαδή τα κράτη θα κάνουν στρατηγικά σχέδια και κάθε κράτος θα έχει διαφορετική στάθμιση και κέντρο βάρους. Για μας όμως παραμένουν οι προκλήσεις για τα αγροκτήματα, το περιβάλλον, το κλίμα, οι αγορές, ε, οι ε, αστάθειες στις αγορές. Θέλουμε τελείως διαφορετικό προσανατολισμό. Όλη αυτή την πρόταση δεν τη θεωρώ καλή αυτή Όπω όπως είπατε στην αρχή, το θεωρώ μια χαμένη ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε τα χρήματα τώρα για να μετασχηματίσουμε ε, τη Γεωργία. Ε, και θα ξαναπώ αυτό που είπε ο Μάρτιν Χόισλινγκ. Πάρτε πίσω ε, την πρόταση, αποσύρετε τη και φέρτε μια καλύτερη. Ευχαριστώ κύριο Χόιτμαν. Στην εισαγωγή σας κύριε Επίτροπε είπατε ότι οι αγρότες εξαρτώνται πάρα πολύ από τη στήριξη του εισοδήματός τους. Γύρω στο 46% έρχεται από τις άμεσες ενισχύσεις από το τις Βρυξέλλε. Αυτό με σόκαρε. Είναι νοσηρό αυτό, δεν είναι υγιέ. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Και η απάντηση δεν είναι να τα αυξήσουμε ακόμα περισσότερο. Θα πρέπει να αυξήσουμε το εισόδημα που μπορεί να πάρει ο αγρότης από την αγορά. Στην πρότασή σας ε, χαίρομαι που εστιάζετε περισσότερο στην αγορά και ε, στην ανταγωνιστικότητα του κλάδου που θέλετε να το δονώσετε παντού στην Ευρώπη. Γενικά χαίρομαι πάρα πολύ με την πρότασή σας. Είναι κομμένη και ραμμένη στα μέτρα των προκλήσεων που θα έχουν στο απότερο μέλλον οι ε, αγρότες και θα είναι και ε, ανταγωνιστική και βιώσιμη γεωργία και όχι με την παλιά παραδοσιακή ε, και παλαιομοδίτικη ε, στήριξη εισοδήματο. Έχω μια ερώτηση. Καμιά φορά ή μάλλον πολλές φορές χρησιμοποιείται με αλφαγιώτα το επιχείρημα ότι χρειάζεται να στηρίξουμε τους αγρότες μας διότι έχουν ανταγωνισμό από τρίτες χώρες. Ο προκάτοχός μου ζήτησε μια μελέτη Έχετε κάνει μελέτες για το κόστος ε, και τη σύγκριση της παραγωγής εδώ με άλλες χώρες ανταγωνίστριες. Ευχαριστώ. Ο πρόεδρος χωρίς μικρόφωνο. E, Είναι σημαντικό και η αγορά να μπορέσει να συμβάλλει. Έχετε δίκιο. Κύριε Επίτροπε, ας το πούμε ειλικρινά, κύριε Επίτροπε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταπιεί κανείς αυτό το προπολογισμό. Το σόκ είναι μεγάλο για τους ε, γεωργούς και πραγματικά φαίνεται ότι υπάρχουν ορισμένα πράγματα που δεν γίνονται κανονικά στις Βρυξέλλες. Τρία χρόνια τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο και η πρότασή σας, η πρόταση της Επιτροπής μάλλον, προτείνει την μείωση της υποστήριξης και την αύξηση ε, η οποία δεν αφορά το γεωργικό εισόδημα. Μπορούν, να, μπορούμε να καταλάβουμε για ποιο λόγο υπήρξαν τόσες επικρίσεις. Παρατήρησα ότι στην ανάλυση δεν λαμβάνεται υπόψη το κόστος του προπολογισμού και δεν λαμβάνεται υπόψη και η εξέλιξη των εμπορικών συμφωνιών. Παρόλα αυτά υπάρχει κάτι σε αυτό που θεωρούσαμε δεδομένο. Η, η, η, πολιτική. Οι γεωργοί δεν θέλουν μια νέα μεταρρύθμιση. Μετά από το σοκ θέτει ο καιρός η σκέψη που είναι αναγκαίος. Θα πρέπει να καταβάλλετε κάθε προσπάθεια, κύριε Επίτροπε, για να μας εξηγήσετε ότι οι προτάσεις που ψηφίστηκαν από το Κοινοβούλιο αναφέρονται και στο κείμενό σας. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ. Ο προϋπολογισμός υποβάλλεται από την Επιτροπή, όχι από τον Επίτροπο Γεωργίας. και οι επικεφαλείς ε, των κρατών θα έχουν άποψη σχετικά με αυτό το θέμα. Ε, Κύριε Σπάης, ευχαριστώ Πρόεδρε. Κοιτάξτε, εμείς οι αγρότες παίρνουμε ένα μεγάλο κλάσμα του εισοδήματός μας από ενισχύσεις αλλά καλύτερα θα θέλαμε να έχουμε τις σωστές τιμές για τα καλά τρόφιμα που παράγουμε και υπό τις συνθήκες που τα κάνουμε. Και θα πρέπει να εξηγούμε όλο και περισσότερο στην κοινωνία γιατί παίρνουμε ενισχύσει και η κοινωνία περιμένει παραγωγή υγιεινών τροφίμων που σεβόμενο το περιβάλλον, γι' αυτό θα πρέπει να στραφεί προς τα εκεί ενίσχυση. Δεύτερον, εγώ καλλιεργώ βιολογικά και πληρώ όλους τους ε, στόχους για το περιβάλλον, για τα νερά, για τα ζώα και ό,τι άλλο θέλουν τα έγγραφά σα. Και πού ε, είναι ο κλάδος μου, είναι περιφθοριακός. Η βιολογική γεωργία υπάρχει ως στόχος για την ε, στήριξη και αν θέλετε να βοηθήσετε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, βάλτε ένα κατόφλι ε, ε, δύο μονάδων μεγάλων ε, ζώων ανά εκτάριο, δύο γυαλιολάδια δηλαδή το εκτάριο, για να μην είμαστε απέναντι στις τεράστιες γιγαντίες εκμεταλλεύσεις των Αμερικανών με τον Αραβόστο και τη Σόγια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε που αναφέρεται τα κυρία στοιχεία της έκθεσης Τόρφων ε, με εξαίρεση του οικονομικού κονδυλίου. Και είναι ένα πολύ άσχημο μήνυμα. Η Επιτροπή Προπολογισμών εξέφρασε την επιθυμία να διατηρηθεί το κονδύλι της κοινή αγροτικής πολιτικής. Θα βρείτε λοιπόν μια υποστήριξη από την Επιτροπή Προπολογισμού, κύριε Επίτροπε. Χαιρετίζω ε, στις προσπάθειες που προτείνεται για την ε, μείωση της πολυπλοκότητας ε, και των διατυπώσεων. Ακόμη και αν έχω κάποιες αμφιβολίες σε σχέση με την αποτελεσματικότητα αυτής της απλούστευσης, όμως σίγουρα αυτό πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα. Έτσι λοιπόν είμαστε στην έναρξη των διαπραγματεύσεων και όρθως υπενθυμίσατε ότι η Γαλλία υποστήριζε το, τα κονδύλια της κοινή γεωργικές πολιτικές. Ε, Μην διστάσετε να πείτε στον κύριο Έτικερ, στον αρμόδιο για τον προπολογισμό, ότι όταν ε, θα μιλήσει στις ε, κοινοβουλευτικές επιτροπές στη Γαλλία για τον προπολογισμό, ότι υπάρχει διπλή γλώσσα Σίγουρα θα κερδίζαμε σε αποτελεσματικότητα και α είμαστε ξεκάθαροι, η κοινή αγροτική πολιτική δεν είναι ένα θέμα ρύθμιση και προπολογισμού, αλλά είναι και ένα θέμα συνοχή μεταξύ τη πολιτική ελεύθερων συναλλαγών και τη ε, πολιτική που έχει να κάνει με την επιστημική ασφάλεια και την κυριαρχία. Θα ήθελα λοιπόν ε, να μπορούσαμε να κάνουμε μια επίσημη διακήρυξη για να πούμε ότι θα υπάρχει μια συνοχή μεταξύ τη κοινή αγροτική πολιτική και τη πολιτική ελεύθερων ε, συναλλαγών. Δηλαδή να μην επιδοτούμε ανθρώπου που θα θέσουμε σε χρεοκοπία ε, για να δεχτούμε συνθήκε εισαγωγών που δεν θα είναι βιώσιμε. Κυρίε και κύριοι, δεν μπορούσα να περιορίσω το χρόνο αγόρευσης ε, του Πρόεδρου Επιτροπής Προπολογισμού, καθώς είναι και αντιπρόσωπος ε, της δικής μας, ε, αντιπρόεδρος, της Επιτροπής, κύριε Ζωάν. Κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ για τις προσπάθειες που κάνατε και είναι προφανές ότι η δουλειά σας προσπαθεί να απαντήσει στα συμφέροντα και τις επιθυμίες όλων των κρατών μελών. Βέβαια, υπάρχουν κάποια πράγματα για τα οποία είμαστε δυσαρεστημένοι και θα θέλαμε να βελτιωθούν. Μιλήσατε για τις επιδοτήσεις. Συμφωνώ που έχετε διατηρήσει και τους δύο πυλώνες, όμως δεν συμφωνώ με τη μείωση του πυλώνα 2. Ωστόσο, εφόσον ε, μιλάμε για επιδοτήσεις, ε, θα ήθελα να μου πείτε και να καταλάβω γιατί εξακολουθούν να υπάρχουν διαφοροποιημένες πληρωμές μεταξύ των γεωργών των κρατών μελών. Ε, γιατί, το χάρη, ένας Γάλλος γεωργός λαμβάνει τα διπλά απέναντι σε ένα Ρουμάνο γεωργό, γιατί τη στιγμή, ε, τη στιγμή μάλλον που υιοθετήθηκε αυτό ήταν διαφορετικό το κόστος. Σήμερα το κόστος είναι το ίδιο και στα δύο κράτη, όμως ε, στα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης έχουμε μεγαλύτερο κόστος παραγωγής γιατί δεν υπάρχει τόσο μεγάλη βιομηχάνηση όπως στα άλλα κράτη. Κύριε ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, κύριε Επίτροπε, είπατε ότι ε, θέλετε κρατικές ενισχύσεις πιο δίκες. Αυτά είναι στα λόγια όμως, γιατί οι συγκεκριμένες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, αντιτίθενται σε αυτό. Έχω την εξή ερώτηση. Αν θέλετε να εφαρμόσετε την αιρεσιμότητα και να εξαρτήσετε τις ενισχύσεις από το κράτος δικαίου, για ποιο λόγο η ίδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην καταβολή των άμεσων ενισχύσεων δεν σέβεται τη συνθήκη προσχώρηση των χωρών που υπέγραψε η ίδια. Πείτε μας σαφώ ποιο είναι το ποσοστό ε, του έσου όρου του ευρωπαϊκού που θα πάρουν οι, Πολωνίοι οι Πολωνοί μάλλον αγρότες. Ε, γίνονται κάποιες αλλαγές, κάποιες μετατροπές. Όλα αυτά έχουν ένα κόστος. Τα έχετε υπολογίσει, έχετε στοιχεία αυτά για το κόστος ε, από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό που πηγαίνει στα κράτη-μέλη. Είπατε ότι το πρασίνισμα είναι αποτυχία και τώρα το έχετε εγκαταλείψει. Ε, εγκαταλείψει. Επίσης δηλώσατε ότι η προστασία του κλίματος είναι κάτι που θα εγκαταλειφθεί. Είναι τελείως παράδοξο όλα αυτά. Η Γεωργία να πρέπει να προστατεύει το κλίμα. Αυτό που λείπει από την πρότασή σας είναι πραγματικά μια υγιής και βιολογική γεωργία. Η κυρία Πετήρ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστούμε που ήρθατε εδώ στην Επιτροπή μας. Σε ό,τι αφορά τη συνθήκη προσχώρησης Κροατίας είχαμε μία μεταβατική περίοδο μέχρι το 2022. Κατά τη διάρκεια της περίοδου αυτής η Γεωργία της Κροατίας ε, θα μπορούσαν να λάβουν ένα μέρος των πληρωμών από τον πρώτο πυλώνα από τον Εθνικό Προϋπολογισμό και ένα τμήμα από το Ταμείο Εγγύσεων η Κροατία έφτασε σε ένα πλήρες ποσοστό πληρωμών το 2020 θα φτάσει και δεδομένου των περικοπών στην ΚΑΠ θα ήθελα να μου πείτε αν η Κροατία θα είναι η μόνη χώρα στην ιστορία που δεν θα λάβει ένα πλήρες ποσό από την Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι όπως είχε οριστεί στη συνθήκη προσχώρησης. Η Κροατία θα πληρώσει όλο το ποσό θα, θα πληρωθεί όλο το ποσό που αναφέρεται στη συνθήκη προσχώρησης και θα βοηθήσει την Κροατία για την αφαίρεση των αρκών. Είναι γεγονός ότι έχει γίνει περικοπή στην χρηματοδότηση της γεωργίας της τάξης του 25%. Πώς θα μεταφραστεί αυτό για τις αγροτικές περιοχές στην Κροατία, δεδομένου ότι έχει εκταμιεύσει το 46% του εθνικού της πολυπολογισμού Κροατία για την αγροτική ανάπτυξη. Κύριε Πίτροπε, εγώ έχω μία θέση και έχω και μία ερώτηση. Καταρχήν, ξέρουμε ότι ο προπολογισμό θα μειωθεί. Όμως, ε, θα ήθελα να σας πω ποια είναι η δική μου ιδέα. Ακούμε εδώ ότι μειώνεται ο προπολογισμό ε, της κοινωνικής πολιτικής λόγω των μεταναστευτικών ροών. Όμως ξέρουμε ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να ε, σταματήσουμε τη ροή των ανθρώπων που εγκαταλείπουν τα χωριά ε, για τις πόλεις. Ε, έτσι λοιπόν θα πρέπει να θέσουμε ένα τέλος σε αυτή την εγκατάλειψη των αγροτικών περιοχών από τον πληθυσμό. Θα ήθελα να μιλήσω για κάτι που συχνά ξεχνιάται, κάτι που αφορά τη μελισσοκομεία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Τι θα κάνετε με αυτό. Η κυρία Κάντεμπαχ, στο άρθρο 7 αναφέρεται τους δείκτες και οι δείκτες που έχουν σχέση με το περιβάλλον και τους ειδικού στόχους δίνανται, αλλά δεν οφείλουν να καλύπτουν παρεμβάσεις ε, κτλ που απορρέουν από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Το άρθρο 11 ορίζει ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να συμπεριλάμβουν στο σύστημα ερησιμότητας στο ε, στρατηγικό ε, σχέδιο για την γεωργία και αναφέρονται αυτά και στο παράρτημα 3 κτλ. Αυτά υπολείπονται των όσων σήμερα ε, ισχύουν. Δεν υπάρχει καμία πρόταση για περιοχές οικολογικού ενδιαφέροντος, ούτε για απαγόρευση χρήσης φυτοφαρμάκων σε οποιαδήποτε γη. Ε, ανησυχούμε πάρα πολύ, ιδιαίτερα για τη διαφύλαξη της ε, ποικιλότητας και των εντόμων που κάνουν την επικονίαση. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, είμαι Γεωργία, Γεωργός, 480 εκατομμύρια ευρώ για το προϋπολογισμό 365 για την πρόταση που μα αποβάλλει σήμερα η Επιτροπή. Η συμβολή της ε, Βρετανίας ε, προτιθέμεται 27 εκατομμύρια. Αν κάνουμε τους υπολογισμούς, φτάνουμε στα 316 ε, δις. Πραγματικά να αναρωτιέμαι. Έχω την εντύπωση ότι το Brexit είναι ένα άλλο τύπο για να μπορέσουμε να καταπιούμε μια μείωση των κονδυλίων του προπολογισμού. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πίτροπε, στην αρχική σας τοποθέτηση τονίσατε ιδιαίτερα τα κοινά της κοινή γεωργικής πολιτικής και είπατε ότι θέλετε να το εγγυηθείτε και στο μέλλον. Διαβάζοντας όμως λεπτομερώς την πρότασή σας βλέπω ότι σε 27 προϊόντα μέχρι και σε 10 ή 13% σε κάποια κράτη-μέλη έχετε συνδεδεμένες ενισχύσεις. Βλέπω ε, να επιτρέπονται πολλές μεταβιβάσεις από τον πρώτο στο δεύτερο πυλώνα και τούμπαλιν. Εάν επίσης ε, δω τι γίνεται στο δεύτερο πυλώνα, μόνο 30% είναι οι ελάχιστες ποσοστώσεις ε, που προτείνεται για την περιβαλλοντική πολιτική και μέχρι και 75% λέτε των επενδύσεων ε, που μπορούν να ενισχύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διερωτώ με ποια είναι τα κοινά και πού είναι τα κοινά. Και στο τέλος μήπως ξαναπέσουμε σε μια επανεθνικοποίηση. Φλάναγκαν. Ο κύριος Φλάναγκαν. Ε, thank you very much. Ευχαριστώ. Πριν από μερικά χρόνια αν κάποιος ε, ε, άκουγε ότι θα γίνει μία ανακοίνωση για την ΚΑΠΑ, θα έλεγε ότι από τη στιγμή που είμαι αστός δεν με ενδιαφέρει, αλλά σήμερα η ΚΑΠΑ σε ενδιαφέρει όλους. Εδώ έχουμε να κάνουμε με μία ληστεία και η Επιτροπή οδηγεί το αυτοκίνητο με το οποίο απομακρύνονται οι ληστές. Ε, δεν μπορεί να γίνει η ανακατανομή ενός πράγματος που δεν υπάρχει. Δεν μένουν πάρα πολλά για να ανακατανείμουμε. Μιλάμε για ε, ε, μεγάλες ε, περικοπές, αν λάβουμε υπόψη ναι, τις περικοπές στην απασχόληση, το όλο θέμα καθίσταται αν, ανούσιο. Υπάρχουν άνθρωποι που υποστηρίζουν ότι είναι γεωργοί, λαμβάνουν 120.000 ευρώ το χρόνο και δεν κάνουν τίποτα. Δεν θα υπάρξει ανακατονομή και θα υπάρξουν βασικές αλλαγές. Δεν βλέπω να υπάρχει καμία σχέση μεταξύ της έκθεσης του κυρίου τόπανα αν συνεχιστεί η κατάσταση. Πώς θα, πώς θα το συνδέσουμε με ανθρώπους και αυτό που έκαναν πριν από 27 χρόνια. Θα πρέπει να μιλήσετε για αυτό που κάνουν οι άνθρωποι αυτό τώρα. Αγνοήσατε πλήρως αυτά που είπαμε. Τελείωσα, Πρόεδρε. Ακούσατε, ε, ακούστε, μιλά, μιλήσατε το διπλό από ό,τι έπρεπε. Έχω μια παρατήρηση και μια ερώτηση. Πρώτα την παρατήρηση. Κύριε Πίτροπε, θέλω να σας πω ειλικρινά ότι δεν το θεωρώ σωστό να έρχεσαι τελευταίο στο κοινοβούλιο. Το έχουν συζητήσει οι βουλευτέ. Πήγατε πρώτα σε όλα τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα. Πρώτα δώσατε συνέντευξη τύπου, τελευταίο το κοινοβούλιο. Δεν είναι καλή εικόνα. Προηγουμένω είπατε τι ωραία που έχουμε εδώ του βουλευτέ. Ε, πρέπει να πω ότι η ευγένεια είναι πιο διαδεδομένη στο Κοινοβούλιο, φαίνεται, από ό,τι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μιλήσατε για ενίσχυση των εργαζομένων. Ε, ε ενώ Ποιοι είναι οι πραγματικοί εργαζόμενοι ή όσοι δηλώνονται αριθμητικά. είναι οι πραγματικοί εργαζόμενοι που πραγματικά δουλεύουν σε μια εκμετάλλευση. Ε, εγώ ενδιαφέρομαι πάρα πολύ ως σοσιαλδημοκράτης ότι θα πρέπει να ενισχύονται εκείνοι που είναι ασφαλισμένοι κανονικά με εισφορές, πληρώνουν φόρους κλπ αυτές οι θέσεις εργασίας. Δεν μπορούμε να μιλάμε για θέσεις εργασίας στη μαύρη αδήλωτες και τέτοια πράγματα. Το ξέρω ότι υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις που προβλέπονται για οικογενειακές εκμεταλλεύσεις. Σωστό είναι αυτό και να το συζητήσουμε. Αλλά ενίσχυση των εργαζομένων από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αφορά μόνο κανονικές θέσεις εργασίας. Ευχαριστώ πολύ. Πράγματι. Πράγματι. Α, συγγνώμη. Πράγματι είναι έτσι τα πράγματα. Μετά τις διαβουλεύσεις μας, οι επίτροποι συζητάνε με τους δημοσιογράφους. Οργανώσαμε τα πράγματα με αυτόν τον τρόπο και ελπίζω ότι τα καταλάβετε. Ο κύριος Κατάινεν. Κυρία. Ε, κύριε είναι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πίτροπο για την παρουσίασή του. Μερικές από τις προτάσεις αντικατοπτρίζουν το πώς οι ευθύνε μετακυλώνται στα κράτη-μέλη. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Παρόλα αυτά, αυτά η αιρεσιμότητα απαιτεί μεγαλύτερη ελαστικότητα. Υπάρχουν ορισμένε περιοχές που δεν έχουν ληφθεί επαρκώς υπόψη. Δεν μπορούμε να δεχτούμε τις περικοπές για αγροτική ανάπτυξη. Σε ό,τι αφορά το κάπινγκ θα πρέπει να ρωτήσω ποιος είναι ο στόχος ε, της Επιτροπής με το ανώτατο όριο. Έγινε μια προσπάθεια να προωθηθεί παραγωγικότητα. Αυτό βεβαίως ε, θα οδηγήσει σε μια μείωση των εσόδων του, του κέρδους για τους γεωργούς. Ευχαριστώ. Αυτό που προκαλεί περισσότερες αμφιβολίες είναι το νέο σύστημα με τα στρατηγικά σχέδια και αν και δεν τον γνωρίζετε υπάρχει κάποιος κίνδυνος επανεθνικοποίησης. Επίσης, η μείωση του προπολογισμού. Το Κοινοβούλιο κατά πλειοψηφία είναι κατά της μείωσης του προπολογισμού. Θέλω να κάνω βέβαια κάποια συγκεκριμένη ερώτηση. Γιατί βγάζετε τον κανονισμό του Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης από τα διαφορετικά ταμεία δεν ξέρω ποιος είναι ο στόχος, όμως ε, αυτό που πιστεύετε είναι ότι δεν θα υπάρχει άνεση χρηματοδότησης όταν έχουμε χώρες στόχου 1 ή αν ε, δεν ε, υπάρχουν κριτήρια ε, αφαίρεσης ε, του Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης από τα διευθυντικά ταμεία. Γιατί στο νέο στόχο δεν αναφέρεται η γυναίκα αγρότης. Ε, η γυναίκα είναι πάρα πολύ σημαντική για την πολιτική της υπαίθρου και πρέπει να αναφέρεται η αγρότησα. Επίσης, αν δεν θα εγκριθεί το πολίτες δημοσιονομικό πλαίσιο, τι θα συμβεί. Η κυρία Σχράιερ πήρε και ευχαριστώ πρόεδρε πολύ. Κύριε Πίτροπε, οι δημοσιογράφοι δεν πήραν απάντηση για το πού θα περικοπούν ε, οι δαπάνες. Παραμένει το ερώτημα πόσα λεφτά θα έχουμε στη διάθεσή μας και πού. Και πολύ συγκεκριμένη ερώτηση. Μιλήσαμε για τον πρώτο πυλώνα και για τον δεύτερο πυλώνα. Μιλήσατε για συμβουλευτικά όργανα, μικρομεσαίες εκμεταλλεύσεις και έρευνα. Μα δεν επιτρέπεται χώρες ε, όπως είναι οι ε, κάτω χώρες ε, που είναι πολύ υπέρ της Ευρώπης να έχουν τεράστιες απαιτήσει. Είπατε ότι σφάξαμε 160.000 αγελάδες και οι αγρότες φτωχεύουν. Πώς μπορείτε να εγγυηθείτε ότι ο αγρότης στην Ολλανδία θα μπορέσει να παραμείνει αγρότης. Κύριε Κούσμιουκ. Ευχαριστώ Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, έχω μια στρατηγική παρατήρηση. Εσείς ε, είπατε ότι θα είχαμε κόστος 12 δισεκατομμύρια ευρώ ε, το χρόνο. Για ποιο λόγο λοιπόν η Κομισιόν έχει προτείνει άλλες προτεραιότητες που κοστίζουν ε, άλλα δισεκατομμύρια και τελικά θα έχουμε περαιτέρω περικοπές στις ευρωπαϊκές πολιτικές ε, είναι ιδιαίτερα μη ιδιαίτερα αυτή η προσέγγιση. Επίσης, ε, αναφέρεται το σύστημα άμεσων πληρωμών στα νέα κράτη-μέλη. Πραγματικά αυτά που λέτε ε, ουσιαστικά δεν έχουν ουσία. τα μεταξύ της περίοδου 2021-2027 αν δεν υπάρχει ε, πραγματική ευθυγράμμιση των πληρωμών ε, τα νέα κράτη-μέλη θα κατηγορήσουν ε, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για εισαγωγή διακρίσεων. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Χαίρομαι που η Κομισιόν αγωνίζεται για μεγαλύτερη σύγκληση αφενός αφετέρου Είμαστε δυσαρεστημένοι γιατί στις ε, χώρες της Βαλτικής ε, και στη Λιθουανία ε, θα έχουμε μόνο το 75% του μέσου όρου. Σύμφωνα με τη συνθήκη προσχώρησή μα, πρέπει να φτάσουμε το μέσο όρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Έπρεπε να τον είχαμε φτάσει ήδη το 2013. Αυτό σημαίνει ότι οι γεωργοί μα ε, είναι καταδικασμένοι να μην εργάζονται με ίσους κανόνες. 53.000 ε, Γεωργίδη έχουν υπογράψει μια αίτηση που ε, εκφράζουν την δυσαρεσκιά τους. Όταν μιλάτε για σύγκληση, όντως το εννοείτε. Εννοείτε ότι θα υπάρξουν πρακτικά μέτρα. Αν ναι, πότε. Γιατί όλες οι χώρες πρέπει να ε, έχουν τους ίδιους κανόνες, το ίδιο σημείο φετηρίας και κατάληξης. Ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε. Η σύγκληση που προτείνεται μειώνει τα χάσματα στις άμεσες πληρωμές πολύ λίγο. Γιατί προτείνεται να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία εξίσωσης το 2022. Δεύτερη ερώτηση, προτείνεται να μειωθούν τα κατόφλια ευελιξίας Πιστεύω ότι το σημερινό κατόφλι ε, μας ε, έχει αποδείξει ότι λειτουργεί σήμερα. Και κάτι ακόμα, οι πληρωμές που σχετίζονται με την παραγωγή. Επίσης, ε, προτείνεται μείωση αυτών των καταφλίων. Ε, σε ό,τι αφορά τώρα τις άμεσες ενισχύσεις, εγώ δεν γνωρίζω καμία ανάλυση που να αποδεικνύει ότι υπάρχει διαστρέβλωση του ανταγωνισμού με το σημερινό επίπεδο πληρωμών. Και τελευταία ερώτηση. Δεν υπάρχει δυνατότητα να αποκλειστούν οι μικρές εκμεταλλεύσεις από την περιβαλλοντική οικολογική αιρεσιμότητα, γιατί δεν νομίζω ότι αυτό θα βοηθήσει τις μικρές εκμεταλλεύσεις. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ντόρφμαν, χωρίς μικρόφωνο. Α, ζητώ συγγνώμη. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Μερικά πράγματα από τις προτάσεις σας μου αρέσουν πολύ, όπως ο προσανατολισμός στην αγορά. Ε, αλλά και η πράσινη αρχιτεκτονική. Είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά. Στην πράξη πρέπει να δούμε μήπως έχουμε προβλήματα στο δεύτερο πυλώνα. Ε, καλά, αυτά θα τα δούμε στις λεπτομέρειες και θα τα λύσουμε στο μέλλον. Ε, όταν πρόκειται για το New Deliver Model, ελπίζω να έχετε δίκιο και να δικαιωθείτε και όλα αυτή η αισιοδοξία σας να ε, εφοδοθεί, αλλά ξέρετε έχω δει τόσα πολλά, έχω γίνει άπιστο στο μα. Πρέπει για να πιστέψω να τα δω αυτά, να βάλω το, το χέρι επί τον τύπο των ήλων, γιατί τα έχουμε ακούσει αυτά ξανά και να βάγει ανοιχτά ε, όλες αυτές οι προσπάθειες. Μέτρησαν οι υπηρεσίες σας ε, τη σύμπτωση της δική μου έκθεσης με τις προτάσεις σας. Είναι πολύ γενναιόδοροι αν βρήκαν 90%. Εγώ τουλάχιστον δεν τα ε, βρήκα αυτά τα 90% από τη δική μου έκθεση στις προτάσεις σας. Ε, στον πρώτο πυλώνα θα επιθυμούσα λίγο περισσότερο θάρρος περισσότερο θάρρος γιατί εκεί είναι οι μεγαλύτερες δαπάνε και όταν είναι λιγότερα τα χρήματα θα πρέπει να σκεφτούμε πού θα τα συγκεντρώσουμε και αυτό το κάπινγκ το ανώτατο όριο που προτείνεται δεν είναι αποτελεσματικό. Τα έχουμε ξαναδεί και αυτά και θα πρέπει να τα βελτιώσουμε. Αλλά και αυτό υπάρχει και το Κοινοβούλιο και θα το κάνουμε τις επόμενες μήνες, τουλάχιστον θα το επιχειρήσουμε. Ο Πρόεδρος, κύριε Ντόρφμαν, κοιτάξτε να δείτε. Ε, ε, σας έκανε ε, μια φιλοφρόνηση ο Επίτροπος ε, για την έκθεσή σας. Ε, κύριος Μπούντα. You next. Ευχαριστώ μετά ο κύριος Μπούντα. Τέσσερις ερωτήσεις. Ε, ΚΑΠ, ε, στην Ευρώπη είναι τόσο διαφορετικά τα πράγματα, αν επιχειρήσετε ε, για την ε, μείωση του ανώτατου ορίου, να τα αφήσετε στα κράτη-μέλη και από το πρώτο εκτάριο μάλιστα, ακριβώς γιατί είναι τελείως διαφορετικές οι συνθήκες. Δεύτερο, ε, στο δεύτερο πυλώνα τι θα γίνει, λέει ο κύριος Γιάρ. Τρίτη ερώτηση. Μου λείπει η παλιά βασική πρημοδότηση, θυμάστε, και μετά ήρθε το πρασίνισμα. Τη χάσαμε αυτή, υπάρχει, έχει διατηρηθεί ή μήπως δεν το διάβασα καλά και μου διέφυγε. Και τέταρτη ερώτηση, άρση της γραφειοκρατίας για τον αγρότη. Ε, θα μπορούσα να πω έτσι ε, ε, με κακεντρέχεια να βάλουμε οροφή και νότα το όριο στους διοικητικούς υπαλλήλους γιατί ε, αυτό χρειάζεται προσοχή και άρση της γραφειοκρατίας. Μπορεί να είναι καλή η ιδέα σας αλλά θα πρέπει να φτάνει και στον τελικό δικαιούχο στον αγρότη που αυτός μας ενδιαφέρει στο κάτω-κάτω και πολιτικά. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα κύριο Μπούντα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εκτιμούμε τις προσπαθίες σας, κύριε Πίτροπε, και της Κομισιόν. Ε, ταυτόχρονα, βέβαια, έχουμε για κάποιες δυσαρέσκειες ε, σε σχέση με τη σύγκληση. Φυσικά και θα θέλαμε να ήταν πολύ πιο γρήγορη και σε ένα κατάλληλο επίπεδο για τα νέα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τα νότατα όρια. Υπάρχουν κράτη-μέλη που έχουν πάρα πολλέ εκμεταλλεύσει, πολύ μεγάλε, ε, πάνω από 3.500 στη Ρουμανία, που έχουν πάνω από 500 εκτάρια εγώ ε, μπορώ να σας πω ότι οι μικροί και μεσαίοι γεωργοί δεν μπορούν να σταθούν στην αγορά χωρίς ενίσχυση. Όμως ε, ε, υπάρχουν και άλλες εκμεταλλεύσεις που δέχονται ενίσχυση πολύ μεγαλύτερες. Τώρα, γιατί συζητάμε πάντα για την ευελιξία σε αυτό το κοινοβούλιο. Ξέρετε, ότι ε, το γεγονός ότι μεταφέρεται πολλές ευθύνες ε, στα κράτη-μέλη δεν ξέρω αν θα φέρει μείωση της γραφειοκρατίας. Ε, θα θέλαμε ή αν θα θέλαμε λιγότερους κανόνες από τις Βρυξέλλες και να μπορούσαμε τότε να μιλήσουμε για πραγματική μείωση της γραφειοκρατίας. Κύριε Ριμπέιρου. Κύριε Επίτροπε, εγώ ανησυχώ πάρα πολύ με την πιθανή απώλεια της αυτονομίας ε, του Ποσέη. Εδώ μπορούμε να έχουμε ουσιαστικά ένα δούριο ύπο, γιατί οι άκρος ακριματισμένες περιοχές ε, ε, στο πώς θα ορίζονται οι ανάγκες του από τα κράτη-μέλη να αφισβητηθεί. Εμείς έχουμε μια σειρά αυτόνομων περιοχών. Από την άλλη, οι Ορισμένε περιοχές ε, ουσιαστικά ποινικοποιούνται επί τρία από την ε, μείωση της ε, ΚΑΠ. Εδώ καταφέρεστε κατά τη απόφαση αυτού του Κοινοβουλίου για το ΠΟΣΕΙ και ο κύριος Ζούνκερ μας εγγυήθηκε ότι θα προστάτευε αυτή τη δέσμη μέτρα. Έχουμε μείωση 20% στην αγροτική ανάπτυξη και έχουμε μείωση 30% στη χρηματοδότηση των κρατών μελών. Υπάρχουν κράτη-μέλη που δεν τα καταφέρνουν. Μιλάμε για εθνικοποίηση. Λοιπόν, οι Γεωργοί ήδη πλήρωσαν την κρίση της αγοράς, πλήρωσαν το ρωσικό μπαρκό και τα προβλήματα ε, με τις ποσοστώσεις του γάλακτος. Τώρα θα πληρώσουν και το Brexit. Ε, ε, ουσιαστικά αυτή είναι η συμπεριφορά σας απέναντι στους Ευρωπαίους Γεωργούς. Κύριε Πίτροπε, κάτι που δεν καταλαβαίνω είναι το εξής. Γιατί κάνετε μια πρόταση που δεν είναι κοινή από αυτό που θεωρούμε σωστό και απαραίτητο, λέει ο κύριος Κάρας. Γιατί είναι αυτός ο αυτοεφνουχισμός στην ίδια την πρόταση. Και μετά θα πρέπει να δικαιολογήσουμε γιατί δεν κάνουμε αυτό που θεωρούμε απαραίτητο ε, και σωστό για να επιτύχουμε τους στόχους μας. Και ρωτώ δεύτερον, στο δεύτερο πυλώνα για την απλούστευση της γραφειοκρατίας. Έχετε κάνει καμιά μελέτη για να μπορούμε να ε, συγκρίνουμε την πραγματικότητα με αυτά που περιμένετε εσείς για τις επιπτώσεις και ποιες είναι οι μεταβατικές διατάξεις και ρυθμίσεις που προβλέπετε. Um, Επίτροπε, είπατε ότι στις Βρυξέλλες ε, δεν θα αναφέρονται στον αριθμό των δέντρων εκτάριων και κατά συνέπεια αυτό δεν ε, θα έχει επιπτώσεις ε, στις άμεσες πληρωμές. Η βασική πράξη δεν αναφέρει κάποιο στοιχείο για τον αριθμό των δέντρων. Μόνο ότι αυτό ηχεί ω βελτίωση. Δεν υπάρχει εγγύηση ότι θα υπάρξει μία αύξηση των δέντρων. Οι γεωργοί θεωρούν, κατά πόσο θα μπορούσε να θεωρηθεί αυτή η περιοχή, περιοχή στην οποία θα μπορούσαν να βοσκήσουν ζώα. Θα μπορούσατε να ένα μήνυμα ότι περισσότερα δέντρα θα μπορούσαν να, να φυτευτούν δίχως αυτό να έχει άμεση επίπτωση στις πληρωμές. Ε? Με αυτόν τον τρόπο οι γεωργοί θα μπορούσαν να διαφοροποιήσουν το εισόδημά τους, να βελτιώσουν το σύστημα και, ε, να ε, βελτιώσουν την βιοποικιλότητα. έχεις Πέντε καλά πράγματα που βλέπω. Πρώτον, έχουμε ένα το, το όριο στις πληρωμές ε, που εφαρμόζεται. Δεύτερον, θετική στάση για τους νέους αγρότες. Τρίτον, ενίσχυση ε, των αγροτών ε, και των εργαζομένων και ενίσχυση των ευφυών χωριών. Ωστόσο υπάρχουν ακόμα κάποια διλήμματα. Πώς είναι δυνατόν με λιγότερα χρήματα και στην ανάπτυξη της υπαίθρου αλλά και στο Ταμείο Συνοχής θα εγγυηθούμε αυτό που θέλουμε και πώς θα το επιτύχουμε. Και μετά τα στρατηγικά σχέδια που καλούνται να εκπονήσουν τα κράτη-μέλη. Ε, μήπως δημιουργήσουν ένα πρόβλημα ε, στη συνέχιση των πληρωμών. Μήπως είναι υπερβολική επιβάρυνση για τα κράτη-μέλη το πρασίνισμα και αυτό θα οδηγήσει σε ανισότητα μεταξύ των κρατών μελών. Κύριε Επίτροπε, η συνδραστική μείωση το κονδυλίο στον δεύτερο πυλώνα μας ε, οδηγεί στο να υιοθετήσουμε μια συγκεκριμένη στάση. Ε, πιστεύουμε ότι θα χρηματοδοτηθεί μια άλλη πολιτική όπως αυτή της διαχείρισης της ε, μετανάστευσης. Αυτό σημαίνει πάρα πολύ μεγάλες απώλειες ο προστατευτισμός των μεγάλων δυνάμεων και, το, και το Farm Bill ε, της Αμερικής δεν αποτελεί έργο του κακού Τράμπα αλλά του ευγενούς Ομπάμα. Ε, αυτό προστατεύει τους ε, Αμερικανούς αγρότες ενώ οι Ευρωπαίοι πέφτουν σαν τις μύγες. Αντί να θεωρήσουμε, να αναζητάμε προσχήματα για τον πρώτο πυλώνα, θα πρέπει να προσαρμοστούμε στις ιδιαιτερότητες των διαφόρων κλάδων. Μόνο με αυτόν τον τρόπο οι χώρες μας θα μπορέσουν να σταθεροποιήσουν τον αριθμό των γεωργών καθώς και το εισόδημά τους. Το νέο μοντέλο παροχών που μας προτείνεται έχει στόχο να αναλάβουν τα κράτη τη μια στρατηγική διαχείριση. Αλλά οι ιδιαιτερότητες των κρατών μελών δεν, ξέρουν, δεν μπορούν να διαφυλαχθούν. Για ποιο λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Θα πρέπει να πω ότι τρέφω πολλές αμφιβολίες για την πρόταση, μόνο ότι μας διαβεβαιώσατε. Εμείς μιλάμε για μια κοινή αγροτική πολιτική. Λέτε ότι η Επιτροπή θα ορίσει τους στόχους και θα αφήσει στα κράτη-μέλη τη δυνατότητα να ορίσουν λεπτομερώς τους κανόνες. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούσαν να προκύψουν διαφορετικοί κανόνες. Κανόνες ε, που οδηγούσαν μια μείωση. <clears throat> Θα δημιουργηθεί ένα ανομοιογενές ευρωπαϊκό σύστημα το οποίο θα δημιουργήσει αθέμητες πρακτικές. Αφού πρέπει να μιλήσουμε για ευελιξία, εντάξει, χρειάζεται όμως μια κοινή διαχείριση, γιατί υπάρχουν πολλές κοινέ δυναμικές. όταν μιλάμε για την κοινή αγροτική πολιτική. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Δόρος. Κύριε κυρία Δόρος. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε, 75% των προϊόντων της Ιρλανδίας πηγαίνουν στη Μεγάλη Βρυτανία. Το 80% του μοσχαρούισκιου κρέατος προς ε, ε, στην εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εσείς όμως συνεχίζετε να στηρίζετε μια πολιτική που καταστρέφει τη βιομηχανία τροφίμων στην Ιρλανδία βάζοντας ε, τους ελέγχους Είμαι σίγουρη ότι αυτό το καταλαβαίνει ένας Ιρλανδός Επίτροπος. Επικρίνεται και η Ιρλανδική κυβέρνηση και η Επιτροπή οι Ιρλανδοί ε, μένουν σε μία διάμεση κατάσταση. Μπορούμε να διαφοροποιήσουμε τις αγορές, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι δεν μπορούμε να υποκαταστήσουμε όλα τα βασικά αγαθά. Αυτό σημαίνει ότι εξαγοράζουμε τις, αγορά, τις αγορές και υποτιμάμε τις τιμές. Εσείς στην παρουσίασή σας μιλήσατε για την επίπτωση των οικονομικών και του Brexit. Αλλά δεν είπατε τίποτα για την διασφάλιση της πρόσβασης στην αγορά στους Ιρλανδούς γεργούς. Και εγώ θα σας έλεγα να σταματήσετε αυτά τα πολιτικά παιχνίδια με τους γεργούς της Βόρειας Ιρλανδίας. Εκτός μικροφώνου. Η κυρία Χάζεκαμπ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πίτροπε, η μεταρρύθμιση νομίζω είναι υπερβολικός χαρακτηρισμός για τα όσα μας προτείνεται. Η ευρωπαϊκή και η ορική πολιτική συνεχίζει την πεπατημένη και πάλι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει αστρονομικό ποσό 265 δισεκατομμύρια για γεωργικές επιδοτήσεις και ένα μεγάλο τμήμα καταλήγει στη μαζική παραγωγή ε, γαλακτοκομικών και κρέατος και κάθε μέρα υποφέρουν τα ζώα σε τεράστιες εκμεταλλεύσεις, σε βάρβαρα σφαγεία, σε ε, απάνθρωπες ε, συνθήκες μεταφοράς. Έχω μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση. Το Κοινοβούλιο επανειλημμένα έχει ζητήσει να σταματήσουν επιδοτήσεις ε, για ε, να ε, εκτρέφονται ζώα με σκοπό αγώνες. Το Κοινοβούλιο ζητάει η κατάσταση επιγόντως να αλλάξει. Και έχω μια σαφή ερώτηση. Τι θα κάνετε στη νέα γεωργική πολιτική να μην υπάρχουν πλέον γεωργικές επιθετήσεις για να κάνετε ε, τέτοιες επιδοτήσεις ε, σε, σε ζώα ε, που τα χρησιμοποιούν ε, για μάχες και με φρικτούς τρόπους και συνθήκες εκτροφής. Σάντος. ο Ευχαριστώ κύριε Πίτροπε. Καθώς δεν έχουμε χρόνο, θα μπω κατευθείαν στο θέμα. Θα ήθελα να δω ποια είναι η θέση της Επιτροπής σε σχέση με το ΠΟΖΕΙ. ο ίδιο ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεσμεύτηκε να μην μειώσει τον προπολογισμό της πολιτικής αυτής. Όταν αυτή η πολιτική αξιολογείται θετικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως σημαντική για να αντιμετωπιστούν συγκεκριμένες προκλήσεις ε, ε, όπως ε, και η διατήρηση της γεωργικής παραγωγής άκρως από μακρισμένες περιοχές. Επίσης, εκφράζω τη δυσαρεσκιά μου σε σχέση με τις περικοπές για την αγροτική ανάπτυξη, γιατί δημιουργεί μεγάλες διαφοροποιήσεις μεταξύ των γεωργών ανά χώρα και ε, σε σχέση με το πως ε, είναι σημαντικό να διατηρηθεί η ακαιρεότητά του, όπως ε, και η βαθμή ελευθερίας στην προσαρμογή των περιφερειακών αναγκαιοτήτων. Και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που είστε ένας άνθρωπος που συμμετέχει συμμετέχει στο διάλογο. Χαίρομαι και για την επίσκεψη στις Ασόρες. Ε, βέβαια, ε, ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε και να διορθώσουμε όσα έχουν ε, όσα, τα σημεία στα οποία υπάρχουν αποκλήσεις. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ που ήρθατε σήμερα στην Επιτροπή μας. Πολύ κριτική ακούσατε ε, και από τα δεξιά και από τα αριστερά. Αυτό είναι καλό σημάδι μάλλον. Είναι καλέ οι προτάσει σα. Έχω μια πολύ συγκεκριμένη σύντομη ερώτηση για τα στρατηγικά σχέδια που είπατε ότι θα πρέπει να εκπονηθούν και να υποβληθούν ανά χώρα. Αλλά το Βέλγιο έχει δύο περιφέρειες ε, που ε, είναι αρμόδιες για την γεωργία. Δεν υπάρχει εθνική γεωργική πολιτική υπουργείο. Τι θα γίνει λοιπόν, δύο σχέδια θα υποβάλουμε ή θα πρέπει να συνεργαστούμε Φλάνδρα και Βαλονία για να υποβάλουμε ένα εθνικό βελγικό σχέδιο για τη γεωργία. Ο πρόεδρος. Μάλιστα. Αυτά που ακούω Ε, ε, λέτε ότι όταν διαμαρτύρονται όλοι και επικρίνουν όλοι σημαίνει ότι είναι καλέ οι διαπραγματεύσει. Έγινε πολύ καλή συζήτηση. Λοιπόν, κύριε και κύριοι, ε, τελειώσανε οι βουλευτές, δεν έχουμε άλλους που να θέλουν να ρωτήσουν και σημαίνει ότι θα πάρει το λόγο ο Επίτροπος για να απαντήσει. Παρακαλώ. Thank you, uh, and... Uh, Ευχαριστώ. Βλέπω ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την πρότασή μας. Θα κάνω ένα γενικό σχόλιο για το ΠΟΣΕΙ. Νομίζω ότι πολλοί το ανέφεραν, κυρίως ε, άνθρωποι που ανησυχούσαν για το 3,9%. Σίγουρα το ότι αναφέρθηκε ο κύριος Γιούκερ σε αυτό ε, στο παρελθόν δεν ήταν κάτι που είχε απολύτως ε, συνειδητοποιήσει. Θα του το αναφέρουμε λοιπόν ε, και θα το εξετάσουμε με τον Αρμόδιο Επίτροπο για τον Προπολογισμό. Είναι τμήμα των ε, προγραμματών που πάγωσε, όπως ε, και άλλα προγράμματα εκτός από τα προγράμματα για τα σχολεία και την πρόθεση. Κατανοώ τις ανησυχίες των συναδέλφων για το πώς έχει, θα τα συζητήσουμε αυτά. Υποστηρίζω, σε είπε ο κύριος Ντεκάστρο, για το πόσο σημαντικό είναι σε θέση να τα καταφέρουν τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό θα χρησιμοποιήσουμε οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους εκ των προτέρων. Το λάθος που κάναμε στο παρελθόν, και νομίζω το έχουμε συζητήσει, Πάολο, ήταν το εξή ότι το να βοηθούμε τα κράτη-μέλη, αφού έχει ολοκληρωθεί η νομοθεσία, είναι πολύ αργά. Δεν ερμηνεύουν την νομοθεσία επικοδομητικά, δηλαδή έτσι ε, όπως ε, θα ήθελε το Κοινοβούλιο να ερμηνευτεί η νομοθεσία. Ας ε, προσπαθήσουμε λοιπόν να κάνουμε τα πράγματα διαφορετικά, ίσως θα λειτουργήσει, ίσως όχι. Θα προσπαθήσουμε πάντως να τα βοηθήσουμε με τα στρατηγικά σχέδια και να κατανοήσουν τι ακριβώς θέλει ο συνομοθέτης εκ των προτέρων και θα μπορέσουμε να τους δώσουμε και κάποιους χρηματοοικονομικούς πόρους. 22 από το 20 εφτα 7 κράτη-μέλη έχουν ε, εκφράσει την υποστήριξη να υπάρχουν απευθείας κονδύλια στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Θα πρέπει να περιμένουμε και θα δούμε. Ξέρετε όμως πώς έχουν τα πράγματα. Χρειάζεται ομοφωνία για να υπάρχουν περισσότερα χρήματα. Και πολλά από τα κράτη-μέλη ε, που τοποθετήθηκαν για τον προπολογισμό είναι πολύ ε, κάθετα για τις νέες πολιτικές προτεραιότητες, άμυνα, τρομοκρατία, μετανάστευση. Ε, ασφάλεια. Υπάρχουν πολιτικέ επιλογέ που πρέπει να γίνουν όταν η Κομισιόν από τον νόμο υποχρεώνεται να παραμείνει εντό των χρηματοοικονομικών παραμέτρων που έχουν προβλεφθεί. Και όπω είπε και ο πρόεδρο τη Επιτροπή Προπολογισμού, αυτή είναι η έναρξη τη διαδικασία και θα προσπαθήσουμε από κοινού να τη βελτιώσουμε και ελπίσουμε ότι θα είναι προ μια θετική κατεύθυνση στον τομέα τη Γεωργία. Αναφέρθηκε ε, συνάδελφος ε, στα εγωπρόβατα, στην κτηνοτροφία. Αυτοί είναι στόχοι που ανήκουν ε, στο μοντέλο υλοποίηση. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να καθορίσουν τις δικές τους προτεραιότητες, το να τους δώσουμε μεγαλύτερη ευελιξία και στην εφαρμογή επιτρέπει στα κράτη-μέλη να ε, μπορούν να έχουν μεγαλύτερη ευελιξία για να αντιμετωπίσουν τα θέματα που τα απασχολούν περισσότερο. Γιατί, ε, παραδείγματο χάρη, ένα γεωργό, ένα κράτο μέλο, διαφέρει το πώ αντιμετωπίζει τα περιβαλλοντικά ε, θέματα ο Έλληνα, παραδείγματο χάρη, από το Δανό. Έτσι λοιπόν ε, θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε και με την ανανέωση της γενιάς των γεωργών να δούμε πώ η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τα κράτη-μελή να κάνει περισσότερα για την ανανέωση της, γενολογική ανανέωση των γεωργών, γιατί είναι πολύ σημαντικό, γιατί θα χάσουν ε, οι αγροτικές περιοχές μα τη ζωτικότητά του. Επίσης, για την κοινωνική συνοχή ε, θέλουμε να τη λάβουμε υπόψη στις συζητήσει μας. Ε, κυρία Χαϊμπατή, ε, τα θέματα Τη διακυβέρνηση, Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και η ΜΚΟ θα πρέπει να την χάνουν διαβούλευση για τα σχέδια, τα στρατηγικά. Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη λοιπόν θα πρέπει να την χάνουν διαβούλευση. Δεν ε, έχουμε αριθμητικά στοιχεία σε σύγκριση με τρίτες χώρες, αλλά ε, και στην περίπτωση που είχαμε αριθμητικά στοιχεία πρέπει να τα ελέγξω ε, με τις αρμόδιες υπηρεσίες μου και ευχαριστώ να σας τα παρουσιάσω αύριο. Μάλλον σκέφτεστε τη Νέα Ζηλανδία. Ε, για το θέμα των άμεσων ε, ενισχύσεων ε, όταν καταργούνται αυτές και ρυθμίζονται όλα από τις αγορές. Όμως υπάρχει εκεί και ένα ισοδύναμο 11 δισεκατομμυρίων ευρώ σε περιβαλλοντικά προβλήματα. Βέβαια, εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να, να αποφύγουμε να γίνουν κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Ο κύριος Νταντέν και άλλοι ανέφεραν τα δημοσιονομικά. Φυσικά είμαστε σε δύσκολη θέση. Είναι χαρτογράφητα νερά όταν ένα μεγάλο μέρος αποφασίζει να φύγει και υπάρχουν και οικονομικές συνέπειες και δεν έχουμε 12 δις από την ΚΑΠ όπω είπε η κυρία από την Ολλανδία, είναι από όλο τον ε, προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι καθαρή συνεισφορά του Ηνωμένου Βασιλείου. Έτσι λοιπόν ε, το μερίδιο των 12 δισεκατομμυρίων ε, είναι ένα μέρο αυτών που αναλογεί στη Γεωργία. Αυτή είναι η καθαρή συνεισφορά που καταβαλόταν στον προπολογισμό τη Ένωση από το Ηνωμένο Βασίλειο. Όμω αυτό μα δείχνει ότι δεν θα είναι εύκολο να το πουλήσουμε αυτό, εκτό αν πάρουμε περισσότερα χρήματα από τα κράτη-μέλη. Και έχω κάποια σχόλια γι' αυτό. Πιστεύω ένθερμα Όπω υπάρχει και στην έκθεση Ντόρφμαν, ε, για την ανάγκη επιστημιστική ασφάλεια. Ε, Πώ ε, θα το κάνετε αυτό με την βιολογική γεωργία ή με την κλασική γεωργία. Αυτό είναι ένα θέμα επιλογή. Υποστηρίζουμε του βιολογικού γεωργού πάρα πολύ στον πυλώνα 2. Όμω, εσεί θέλετε να έχουμε αποκλειστικά βιολογική γεωργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοιτάξτε, είστε πολύ γενναιόδοροι, αλλά να βολευτείτε με κάτι λιγότερο. θα πρέπει να βασιστούμε σε κάποιου συγκεκριμένου κανόνε και πρόσφατα αναθεωρήσουμε, αναθεωρήσαμε τον κανονισμό για τη βιολογική γεωργία ε, και θέλουμε ουσιαστικά να σεβόμαστε λίγο περισσότερο το τι σημαίνει όρος βιολογικός. Καλωσορίζω το όσα είπε πρόεδρος ε, της Επιτροπής Προπολογισμού για την ανάγκη περισσότερη χρηματοδοτική υποστήριξη από τον προπολογισμό. Πιστεύει ότι θα πρέπει να υποστηριχθεί η ΚΑΠ και αυτό είναι πολύ καλό να το ακούμε από τον πρόεδρο τη Επιτροπή Προπολογισμού. Το καλωσορίζουμε. Όμω, αν ε, είχαμε περισσότερε ε, άμεσε ενισχύσει, θα συμφωνήσετε ότι θα είχαμε πολύ μεγάλη δυσκολία να το ξαναβάλουμε αυτά τα χρήματα στον πυλώνα 1 παρά στον πυλώνα 2, γιατί έχουμε επιλογέ στον πυλώνα 2 και θέλουμε να έχουμε ίσους κανόνες και στις πληρωμές του πυλώνα 1, όμως τα κράτη-μέλη μπορούν να βάλουν περισσότερα χρήματα στον προπολογισμό και μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν για τον πυλώνα 1 ή τον πυλώνα 2, ενώ τα κράτη-μέλη μπορούν να βάλουν ε, απευθείας περισσότερα κονδύλια για τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης. Έχουμε την επιλογή 15% σε κάθε κατεύθυνση. Αν επιπρόσθετο 15% μεταφέρεται από τον πυλώνα 1 στο 2 χωρίς συγνατοδότηση, πρέπει να αφορά περιβαλλοντική δράση και εγκληματολογική δράση και για την ε, εμπορική πολιτική. Συμφωνώ, θα πρέπει να εξετάσουμε το θέμα της εμπορικής πολιτικής, ε, όχι ξέχωρα από το τι κάνουμε, αλλά για να δούμε ποιος θα είναι ο αντίκτυπος στην Ευρωπαϊκή Γεωργία. Και υπάρχουν ευαίσθητα σημεία. Ε, φυσικά έχει ρόλο το Κοινοβούλιο, αλλά και τα κρατημέλη έχουν ρόλο να παίξουν. Είχαμε μάλιστα και την, ε, ε, τον αρμόδιο που πήγε στην Αυστραλία και ενυπομονούσε να ανακοινώσει τη Συμφωνία Αυστραλίας-Νέα Ζηλανδία. Η κυρία Μάλστρομ. Η κυρία Ζωάννα αναφέρθηκε στην εξωτερική σύγκληση. Μπορούμε να κάνουμε περισσότερα εδώ, ίσως. Όμω, ε, ποιε απαιτήσει έχουμε για τον προπολογισμό. Μπορούμε να κάνουμε πολλά. Ακούσαμε και για το ΠΟΖΕΙ τελικά πρέπει να δούμε πώς θα διεξαχθούν οι διαπραγματεύσεις. Ε, όμως, ε, ουσιαστικά, έχουμε πολλές χώρες που έχουν σημειώσει πρόοδο στην Ανατολή. Στη Λιτουανία είχαμε αύξηση 4,2%, ενώ όλοι ταυτόχρονα έχουν μείωση 4% σε σχέση με την ε, στήριξη ΚΑΠ στον πυλώνα 1. Εστονία, Πορτογαλία επίσης έχει λίγο φελθεί. Δεν σας άκουσα να το αναφέρατε αυτό, ούτε αναφέρατε τα 9 εκατομμύρια που πήρατε στη Λιθουανία για τις πλημμύρες. Από την πολιτική της ΚΑΠΡΟ έρχονται αυτά. Και προσπαθήσαμε να αντικατοπτρίσουμε ε, τα προβλήματα, συγγνώμη, να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα με το ρωσικό εμπάργκο. Είχαμε 1,5 δις Προσπαθήσαμε να έχουμε τα απαραίτητα χρήματα από είναι Επιτροπή Προπολογισμού και μπορέσαμε να κάνουμε κάτι για να βοηθήσουμε του αγρότε μα. Ποτέ δεν θα αρκεί αυτό, αλλά υπάρχει ουσιαστικά η αναγνώριση ότι είχαμε ένα πρόβλημα και είχαμε ιδιωτική μαθηματοποίηση ε, στη δημόσια παρέμβαση για να, να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους γεωργού μας. Και πολλοί από αυτούς τους γεωργού επιβίωσαν από αυτούς τους δύσκολους καιρού, ιδίω το 2015 ενισχύσεις που ε, συνδέονται επιδοτήσεις με το κράτος δικαίου. Δεν ξέρω τη θέση της Πολωνίας. Αυτή είναι μια μεγάλη συζήτηση. Η σημερινή αρχιτεκτονική για το πρασινισμό αντικαθίσταται από άλλη περιβαλλοντική και κλιματική δράση. Δεν το καταργούμε αυτό το πράσινο σκέλος, αλλά το, το κάνουμε διαφορετικά και πιο φιλόδοξα και λιγότερο περίπλοκο. Βεβαίω είμαστε πιο φιλόδοξοι και το κάνουμε διαφορετικά. Όλε οι εκθέσει που διαβάζετε, ιδιαίτερα του ελεγκτικού συνεδρίου, μα έχουν πει ότι η σημερινή πολιτική δεν αποδίδει ε, ω προ τη φιλοδοξία μα για το περιβάλλον. Κυρία ε, Πετήρ, η συμφωνία προσχώρηση τη ε, Κροατία γίνεται πλήρω σεβαστή για το 2022. Κύριε Νέκοφ, είχαμε αυτή τη συζήτηση στη Βουλγαρία πρόσφατα θα πρέπει να είναι ομόφωνη η απόφαση. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να συνεισφέρουν για να ε, είναι όλοι ικανοποιημένοι σε ένα φιλόδοξο προπολογισμό. Και κάποια κράτη-μέλη δεν θέλουν να συνεισφέρουν περισσότερο και κάποια άλλα δεν θέλουν να παίρνουν λιγότερα. Ε, τετραγωνισμό του κύκλου. Για να δούμε. Τα έχουμε ξαναδεί πολλές φορές. Τώρα όμως έχουμε ιδιαίτερο ορισμό για ε, τα έξυπνα χωριά. Τα είπαν ο κύριος Σάνη και ο κύριο Μπόκοβιτς και δεν έχουν σχάσει καθόλου τις μέλησης. Ε, θα γίνει και μια πρόταση για την επικονίαση ξεχωριστά ε, για να δούμε πόσο μεγάλη σημασία έχουν οι μέλησεις για τη γεωργία. Αλλά αυξάνουμε τον προπολογισμό για τη μελισσοκομεία από 47 εκατομμύρια ευρώ που είναι πολύ περιορισμένα σε 60 εκατομμύρια. Ε, τουλάχιστον αυτό το μικρό έχει γίνει. Και να πω και στην κυρία Κάντενμπαχ ότι θα κάνουμε πρόσφατα πρόταση για τα έντομα που κάνουν την επικονίαση. Την ξέρετε τη θέση μου για αυτά τα θέματα. Και, και η κυρία Νόιχελ, θυμάμαι το είχε κάνει. Ε, σε σχέση με τόσα είπε η κυρία Ντελαέ και τα στοιχεία που έδωσε. Η ε, Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 έχουν 382 ε, δις. 410 ήταν μαζί με το Ηνωμένο Βασίλειο. 382 για τα 27 κράτη-μέλη. 3,65 είναι σήμερα. Και μετά ε, η συγχρηματοδότηση έχει μειωθεί κατά 10 ποσοστιαίες, όχι 10 ποσοστιαίες μονάδες. Περικοπή ε, ε, οριζόντια. Είναι 10 κάτω. Ε, δεν είναι ποσοστίε μονάδες, είναι εκατομμύρια. Ε, δισεκατομμύρια. Από τα 53 στα 43. Και θα πρέπει να επανέλθει αυτή η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για το δεύτερο πυλώνα. Κύριε Λίντ, πού το βρήκατε το 65% των επενδύσεων που πάει στο δεύτερο πυλώνα. Δεν ξέρω, μήπως θα μου πείτε μετά. Δεν το καταλαβαίνω. Το, πού το βρήκα το 65%. Δεν το έχω ξανακούσει αυτό το στοιχείο. Αλλά μήπως το έχω μπερδέψει. Η εθελοντική υποστήριξη της οροφής, η Γερμανία, ε, είναι αντίθετη ε, σε όλα αυτά. Όχι σε όλα. Εσείς έχετε την πολυτέλεια να εκπροσωπείτε τη Γερμανία. Εγώ θα πρέπει να μιλήσω για 27 ε, κράτη-μέλη. Έχουμε μειώσει στο 10% την πρόταση, αλλά επιτρέπουμε και 2% ε, για κάποιες καλλιέργειες που σας ενδιαφέρουν και σας. Αλλά και πάλι αυτό είναι τα πρωτεϊνούχα φυτά. Κύριε Φλάναγκαν. Πραγματικά με εξέπληξαν τα όσα είπατε. Δεν με εξέπληξαν. Αν το κάπνινγκ δεν δημιουργεί χρήματα, εναπόκειται στι χώρες μέλη να τα ρυθμίσουν αυτά τα θέματα. Θα πρέπει να αποφασίσουν το σύστημα ανακατανομών. Θέλετε να γνωρίζετε πώς μπορεί να γίνει αυτό, έτσι ώστε να είναι υπέρ των μικρών ε, εκμεταλλεύσεων. Βεβαίως υπάρχει πεδίο εδώ εφαρμογής ε, της πρότασης. Ε, αρκετές φορές το έχω τονίσει αυτό. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε. Και βεβαίω αν έχετε τροπολογίες καλείστε να τις υποβάλλετε. Κυρία αυτή είναι η πρώτη ευκαιρία που δεν ε, ελεύθερη η Επιτροπή δεν θέλω να δείξω έδαψη έλλειψη σεβασμού. Ακούσατε τον πρόεδρο να σας εξηγεί πώς ακριβώς ε, έγιναν τα πράγματα. Το Omnibus ασχολήθηκε με μια σειρά από θέματα και όλοι συνέβαλαν σε αυτό. Δεν είναι εύκολο αυτό το θέμα. Υπάρχουν ε, λύσεις διαφορετικές για τα διαφορετικά κράτη-μέλη θα... ήθελα πραγματικά αν είναι δυνατόν το 100%, της, ε, το 100 της ενίσχυσης να καταλήξει στα χέρια των ε, γεωργών. Εγώ βεβαίω δεν μπορώ να κάνω πάρα πολλά για το σύστημα φορολόγησης. Εάν βεβαίω υπάρχει κάποιο πρόβλημα μπορούμε να, να κάνουμε μία αναφορά στην όλα. Ε, η, Φιλα... η Φιλανδία έχει μεγαλύτερη ελαστικότητα σε ό,τι αφορά τον ε, πυλώνα 2. Το αναφέραμε αυτό το θέμα. Αναφερθήκατε στην ε, στήριξη και την αντιμετώπιση κλιματολογικών προβλημάτων. Έγινε μία άλλη αναφορά και θα ήθελα να σας ε, διαβεβαιώσω ότι θα κινηθούμε προς την κατεύθυνση που αναφέρατε. Ε, ε, αν, υπάρχει, αν είναι πρόβλημα της Ισπανίας, δίχως άλλο στο μέλλον θα μας απασχολήσει. Μου λέει ο πρόεδρος ότι θα πρέπει σιγά σιγά να τελειώνουμε απλοποίηση. Θα, πρέπει, ε, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να απλοποιήσουμε τα πράγματα για τον ε, Γιώργο. Ο κύριος Φενόσκι αναφέρθηκε στο 2022. Είναι το πρώτο οικονομικό έτος. Εξαρτάται από τη διαδικασία. Μπορεί να είναι και 2023 ή 2022. Είναι ενδεικτικά ο πρώτος κόνος και θα υπάρχουν εξαιρέσεις ε, για τους μικρούς γεωργούς. Οι χώρες μέλη θα θέσουν ε, στόχους. Ο ε, κύριος Τάτσερ αναφέρθηκε σε αυτό το θέμα του πολιετούς ε, πλαισίου. Η δασοπονία, όπως είπατε και εσείς, ε, θα παίξει καθοριστικό ρόλο, κυρίως σε ό,τι αφορά το κλίμα. Ελπίζουμε να υποβληθούν προτάσεις που θα λαμβάνουν υπόψη τους αυτό το θέμα. Έχω ένα λεπτό ακόμα στη διάθεσή μου. Εγώ δεν βρίσκομαι εδώ για να διαπραγματευτώ το θέμα του Brexit. Νομίζω ότι έχετε πάρα πολλές ευκαιρίες για να το κάνετε αυτό. Ε, γνωρίζουμε το θέμα με τους ε, Ιρλανδούς γεωργούς. Ε, έχουμε τα υψηλότερα δυνατά επίπεδα σε ό,τι αφορά την ευημερία των ζώων. Και η υγεία των ζώων, όπως και η υγεία των ανθρώπων, είναι θέματα που μας απασχολούν. Αυτός είναι ένας από τους συγκεκριμένους στόχους. Η θέση του Βελγίου θα ληφθεί υπόψη στην πρόταση, το γνωρίζουμε αυτό, η συνταγματική θέση και πολλών άλλων χωρών ε, θα ληφθεί υπόψη και αυτό με τις δυσκολίες και στην Ισπανία. Είναι ευαίσθητα θέματα που θα πρέπει να μας απασχολήσουν στην τελική πρόταση. Γνωρίζω ότι δεν απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις, ελπίζω να απάντησα στις περισσότερες. Ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Πιστεύω ότι το πιο δυνατό σημείο είναι τα εργαλεία επίλυσης των κρίσεων για την ε, ε, εξάλληψη της. Πώς θα το λύσουμε αυτό, θα δούμε. Λόγω της ε, διαμάχης με τη διοίκηση δεν θα υπάρξει υπέρβαση ωραρίου. Οι διερμηνεί σα πληροφορούν με τα λήψη ότι συνεχίζεται η εργασιακή διαμάχη με τη διοίκηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τι νέε συνθήκε εργασία. Δυστυχώ, λόγω εργασιακή διαμάχη, η διερμηνία σταματάει τώρα. No, no. Okay. We should, uh, uh, Dziękujemy bardzo. Thank you very much. And e, now it's time for our committee. It's time for our reporters.